Καλημέρα σας. Πάλι σε άλλη αίθουσα πήγα σήμερα. No, θα σου thing you repeat. όχι, όχι, δεν, δεν ξαναλέγονται αυτά. Περνάμε στην ίδια διάταξη. Έχουμε λοιπόν μια αλλαγή της ημερήσιας διάταξης. Η έκθεση Kaiser θα πάει στις 5.30 ώρα. Ε, ξέρω πως δεν χαίρεται ιδιαίτερα η κυρία Λούνατσεκ. Αλλά επειδή είναι νομοθετικό το θέμα, έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Ε, με συγχωρείτε, έτσι πρέπει να γίνει. Ελπίζω να συμφωνείτε. Σήμερα δυόμιση με έχουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Νοτιού Σουδάν. Προσπαθήστε να έρθετε παρακαλώ γιατί νομίζω πως είναι κάτι το σημαντικό αν δει κανείς ότι γίνεται στο Νότιο Σουδάν και το ότι υπάρχει βία. Νομίζω μισή ώρα αξίζει τον κόπο. για την γνωμοδότηση Παλέκης και ανταλλαγή ε, ενεργειακής πολιτικής ε, με τους εταίρους μας. Η προθεσμία για τροπολογία είναι Δευτέρα 26 Μαρτίου. Συμφωνείτε? Ωραία. Έχουμε έξι πρακτικά να εγκρίνουμε. Είμαι σίγουρος ότι τα έχετε διαβάσει όλα. Οπότε υποθέτω πως εγκρίνονται εάν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Παρακαλώ. Περνάμε στον κύριο Κόβατσεφ, το Κόβατσοφ. Θα ε, wird ε, τι έγινε με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας στο Νότιο Κάφκασο, Αζερβαϊτζάν και Αρμενία νομίζω λογικό είναι να το παρουσιάσουμε. Γιατί αύριο έχουμε και το ψήφισμά μας. Έχετε τον λόγο λοιπόν κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα συνάδελφοι. Ε, πολύ ε, χαίρομαι που ένα μήνα μετά την επίσκεψη αυτή στο Αζερβαϊτζάν και λίγο πριν τη συζήτηση για τη Συμφωνία Σύνδεσης ε, με το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία θα ενημερωθούμε για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας στις χώρες αυτές. Ε, ήταν πενταμελή η αντιπροσωπεία, ήμουν εγώ, η κυρία Μακοβέη, ο κύριος Κυρίλοφ, ο κύριος Λάιν και η κυρία Λούνατσεκ. Από 19 μέχρι 21 Φεβρουαρίου. Επίσκεψη στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Με μια στάση στο Γέρεβαν ε, και το, την τυφλίδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και να ευχαριστήσω φυσικά και τη γραμματεία και το προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη. Πριν σας αναλύσω το πρόγραμμα των επισκέψεών μας, να σας παρουσιάσω τα δύο βασικά συμπεράσματα της αντιπροσωπείας. Είναι σημαντική ε, η επίσκεψη αυτή και μάλιστα ο συνδυασμός στις δύο χώρες μαζί με τις παράλληλες συναντήσεις που είχαμε και που έδειξαν τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, τις ημερείς του σχέσεις και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη στάση στην Τυφλίδα ολοκληρώσαμε την ε, εικόνα μας για την περιοχή και υπάρχουν σημαντικές διαφορές ό,τι αφορά τη συνεργασία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν και τη σχέση των δύο επικεφαλής αντιπροσωπιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόθεση της αντιπροσωπείας μας ήταν από την αρχή να ξεπεράσει τη γραμμή επαφών μεταξύ του Αζερβαϊτζάν και του Ορεινού Καραμπάχ, του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Γιατί μετά τη δήλωση του Σότσι πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ε, διατρανώνει τη θέλησή μας για ε, εντονότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην διευθέτηση, στο διακανονισμό του, ορεινού, του προβλήματος του ορεινού Καραμπάχ. Εξαιτής της κακοκαιρίας όμως του χειμώνα, αλλά και επειδή έπρεπε να πάμε με λεωφορείο και δεν υπήρχε και η ε, προθυμία της Αρμενίας να μας ε, διευκολύνει. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε τελικά εκεί. Αυτή η γραμμή είναι πολύ επικίνδυνη, ίσως από τις πιο επικίνδυνες γραμμές ε, του μετόπου σε περιοχές του κόσμου που υπάρχουν τέτοιες διαμάχες. Πάντως, Μετά από αυτά που άκουσα μετά το Συμβούλιο της 27ης ε, Φεβρουαρίου και την πρόθεση για αν επιφύλακτη ανεφόρον πρόσβαση σε όλους τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, θεωρώ ότι είναι θετικά και μου δημιουργώ μια αισιοδοξία. Περιμένω και μια δήλωση από την Αρμενία και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πολύ σύντομα για την ανεφόρον πρόσβαση. Και ελπίζω να συμφωνήσει και η Ερμενία με αυτή την ανεφόρον πρόσβαση. Α, φυσικά και το Αζερμπαϊτζάν. Με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις ε, της α, ε, της ομάδας του Μίνσκ για τον τρόπο διέλευσης αυτής της ε, γραμμής. Πάντως η δική μας απόπειρα έχει και μια θετική επίπτωση. Δεν αναβλήθηκε ή μάλλον δεν απαγορεύεται αυτή, απλώς αναβλήθηκε για το μέλλον. Ελπίζω στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε αυτή την γραμμή διαμάχης. Ε, επισκεφθήκαμε και τον Πακού. Η πρώτη μας συνεδρία στον Πακού ήταν με τον πρόεδρο Αλίεφ. Πριν όμως σας ενημερώσω για τα διαμεθέντα με τον πρόεδρο Αλίεφ, θα ήθελα να θίξω ορισμένα ζητήματα για το Αζερβαϊτζάν. Ε, υπάρχουν αδυναμίες στο πολιτικό σύστημα. Βέβαια, σε, ε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καταρτίστηκαν κάποια σημαντικά νομοσχέδια, αλλά δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή. Ε, δεν, υπάρχει, δεν επικρατεί κράτος δικαίου, περιορισμένες είναι οι δημοκρατικές προδιαγραφές, υπάρχει ενδημική διαφθορά και έλλειψη διαφάνειας σε ό,τι αφορά την, ε, την ε, χρησιμοποίηση των εσόδων από το φυσικό αέριο. Ε, δεν υπάρχουν ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, δεν υπάρχει πρόσφορο κλίμα για την ανάπτυξη της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Από αυτή την άποψη ο διαγωνισμός της Eurovision θα ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για το Αζερβαϊτζάν και ίσως ε, πνεύσει ένας άνεμος εξυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού. Λυπούμε όμως για την απόφαση της αρμενικής τηλεόρασης να μποϊκοτάρει το διαγωνισμό της Eurovision στην, ε, στο Αζερβαϊτζάν γιατί παρά την εξασφάλιση του Αζερβαϊτζάν... Ε, για την προστασία της ε, αρμενικής αποστολής. Λυπούμαστε ειλικρινά για την απόφαση της αρμενικής ε, αντιπροσωπείας να μην μεταβεί στον Πακού και να μην συμμετέχει στο διαγωνισμό της Eurovision. Παρόλο που θα ήταν ένα σημαντικό μέτρο οικοδόμηση εμπιστοσύνη αυτή η συμμετοχή και παρά τι εγγυήσει που έλαβε η Αρμενία από το Αζερβαϊτζάν. Λυπούμαστε ειλικρινά. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνάντηση με τον πρόεδρο Αλίεφ. Ο πρόεδρος Αλίεφ μας ε, εξήγησε ρητά και κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν δεν είναι πολύ πρόθυμη ε, να προωθήσει μια συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτιμά μια στρατηγική εταιρική σχέση σε κάποιες τομείς ε, κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι διαφοροποίηση της προμήθειας, ενεργειακός ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού και επίση ε, υπογράμμισε το ρόλο του Αζερβαϊτζάν στο διεθνέ προσκήνιο, μη μόνιμα μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ και μάλιστα θα αναλάβει και την Προεδρία του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας. Μάλιστα το Αζερβαϊτζάν είναι η, πρώην, ε, ε η μόνη πρώην δημοκρατία της, ε, της Σοβιετικής Ένωσης που προσκλήθηκε στο Μεξικό. βέβαια ε, θέλει να διαδραματίσει πολύ με μετριοπαθή ρόλο στην περιοχή, ε, εξισορροπητικό, έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ και το Ιράν και μάλιστα είναι ένα κοσμικό κράτος μουσουλμανικής θρησκείας και αποτελεί ένα υπόδειγμα, ένα πρότυπο για την περιοχή καθώς και ε, έναν αξιόπιστο ενεργειακό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι φορά τον Αγκόρνο Καραμπάχ, ο πρόεδρος Αλή εφτάχτηκε υπέρ μιας αντικατάστασης ε, της Γαλλίας ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ομάδα του Μίνσκ και περιμένουμε ε, και τη θέση της Ρωσίας εδώ. Είπε πάντως ο πρόεδρος Αλίεφ ότι ο χρόνος είναι με την πλευρά της Αρμενίας ό,τι αφορά την διαθέτηση της σύγκρουσης αυτής. Επίσης είπε ότι η αποτυχία της συνεδρίασης του Καζάν οφειλόταν στις τροπολογίες που τελευταία στιγμή υπέβαλε η Ρωσική Ομοσπονδία. Υπήρχε σαφής διαφορά μεταξύ της ερμηνείας που δίνει η Αρμενία στην αποτυχία της συνάντησης του Καζάν και στην ερμηνεία που δίνει το Αζερμπαϊτζάν σε αυτή την αποτυχία. Και στο Σότσι ο πρόεδρος Αλίεφ είπε ότι, είπε ότι ή μάλλον για το Σότσι είπε ότι ήταν περισσότερο ένας αποχαιρετισμός του Προέδρου Μετβέντεφ η συνάντηση αυτή. Και δεν θεωρεί ότι η διακήρυξη του Σότσι έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ε, θετικές εξελίξεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. συνέχεια, συναντηθήκαμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ασίμοφ, που επέκρινε την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τις συμφωνίες σύνδεσης και πέριψε όλες τις τροπολογίες σε σχέση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμφώνησαν 27 χώρες μέλη. Είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα μοντέλο ενιαίο για όλες τις χώρες. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε συμφωνία σύνδεσης να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Γιατί άλλο, άλλα χαρακτηριστικά έχει το Αζερβαϊτζάν και άλλα η Ουκρανία ή η Μολδαβία για παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά την Αρμενία. Πετάξαμε από τον Πακού στη Διφλίδα και κατόπιν πήγαμε οδικός στο Ερεβάν. πέντε ώρες διήρκησε η διαδρομή με το λεωφορείο, αλλά ήταν ε, η συντομότερη διαδρομή. Ε, μια και δεν μπορούσαμε να περάσουμε τη γραμμή του Ναγκόνο Καραμπάχα, αλλιώς θα χρειαζόταν δεκάωρη, δωδεκάωρη ε, οδική μεταφορά, εκτός αν χρησιμοποιηθεί ελικόπτερο ή κάποιο άλλο μέσο. Πάντως με λεωφορείο θα κρατήσει 10-12 ώρες. Στην πρώτη μας συνεδρίαση με το Γερεβάν συναντήσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών. Ε, θέμα της συζήτησης ήταν κυρίως ε, η κατάσταση στον Αγκόνο Καραμπάχ. Ε, υιοθέτησε ο Υπουργός μια νομικήστικη μάλλον προσέγγιση ως προς τη σύγκρουση αυτή. Είπε ότι θα πρέπει το Αζερβαϊτζάν να επιδείξει κάποιο σεβασμό και δεν θεωρεί ότι η διέλευση της γραμμής επαφής είναι μέτρο οικοδόμηση εμπιστοσύνης. μετά και την τελική διακήρυξη του Σότσι. Επίσης, μας εξήγησε την ε, ε, αρμενική ερμηνεία για την αποτυχία του Καζάν, που όπως σας είπα διέφερε ριζικά από την ερμηνεία του Αζερβαϊτζάν για την αποτυχία της συνάντησης του Καζάν. Και στα συμπεράσματα που θα σας προτείνουμε είναι να συναντήσουμε τον συμπρόεδρο της ομάδας του Μίνσκ, ε, να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί του, γιατί μας ενδιαφέρει και η άποψη του συμπροέδρου της ομάδας του Μίνσκ και την αποτυχία της συνάντησης του Καζάν. Γιατί επαναλαμβάνω ήταν διαμετρικά αντίθετες οι ερμηνείες που έδωσαν το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία για την αποτυχία αυτή. Αυτή θα ήταν μία από τις συστάσεις μας μετά την αποστολή μας να γίνει ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας με τον συμπρόεδρο της ομάδας του Μίνσκ. Συναντηθήκαμε και με τον πρόεδρο Σαρκισιάν. Η συνάντηση ήταν πολύ ανοιχτή, επικοδομητική και καρποφόρα. Ένα μεγάλο τμήμα της αφιερώθηκε και πάλι στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ο πρόεδρος Σαρκισιάν μίλησε για το ρόλο της ομάδας ε, ΟΑΣΕ και Μίνσκ και μίλησε για την αντικατάσταση της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε ότι η διέλευση τη γραμμή επαφή θα πρέπει να... Για να γίνει αυτή η διέλευση θα πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες με τις αρχές των Αγκόνο Καραμπάχ. Πάντως τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται ότι υπήρχε μια μετακίνηση της Αρμενίας ως προς την κατάσταση αυτή, ως προς το θέμα αυτό και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και εξελίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης, συναντήσαμε τον Υφυπουργό Νάστα Κασνιάν, που είναι και επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συμφωνία Σύνδεσης. Μίλησε για πολιτική συνένεση όλων των πολιτικών παρατάξεων της Αρμενίας υπέρ μια σύγκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, μια θετική στάση και της κοινή γνώμης υπέρ της προσέγγιση αυτή. Στα τέλη Φεβρουαρίου 22 από τα 28 κεφάλαια της Συμφωνίας Σύνδεσης έχουν ολοκληρωθεί και μάλιστα ε, ξεκίνησε η σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με την ε, Αρμενία και η Συμφωνία για τη Διευκόλυνση των Θεωρήσεων και ε, τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Τέλος, ό,τι αφορά τις συναντήσεις με προσώπους διεθνών οργανώσεων, think tanks και κοινωνίας των πολιτών, θα ήθελα να υπογραμμίσω την δυσπιστία που υπάρχει μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευσης η οικονομική κατάσταση είναι δεινή, δεν υπάρχουν επενδύσεις, μεγάλη ενεργεία, ε, αυξημένη μετανάστευση, αποδημία μάλλον και ελάχιστες προοπτικές για τους νέους στην Αρμενία. Στις 6 Μαΐου θα διοργανωθούν εκλογές. Θα είναι σημαντική η λιδία για το νέο εκλογικό νόμο της Αρμενίας, γιατί ε, η περιορισμένη ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας ε, είναι γνωστή και υπογραμμίστηκε και στις επαφές μας. Ε, θα είναι πολύ σημαντική η στιγμή των εκλογών ε, στην Αρμενία. Θα πρέπει να είναι δίκαιες, διαφανείς, ανώθευτες, γιατί θα κριθεί η Αρμενία από τις εκλογές αυτές. Και δύο λόγια για τη Γεωργία. Στην Τυφλίδα είχαμε το απόγευμα την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον πρέσβη Φιλίπ Δημητρόφ, και τον ε, ε, αντιπρόεδρο της ε, αποστολής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία. Ήταν μάλλον θετική εικόνα που μας έδωσε ο πρέσβης για τον εξυγχρονισμό της Γεωργίας και ο αναπληρωτής αρχηγός της, της αποστολής παρακολούθησης μας μίλησε για τον μηχανισμό πρόληψης προβλημάτων και τα ζητήματα της Απχαζίας. Πάντως, στόχος ε, της αποστολής αυτής δεν ήταν η κατάσταση στη Γεωργία, αλλά περισσότερο επίσκεψη στο Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Τα συμπεράσματα τώρα. Ήταν πολύ χρήσιμος αυτός ο συνδυασμός των δύο επισκέψεων και οι παράλληλες συναντήσεις και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και με εκπροσώπους της κυβέρνησης, ιδιαίτερα οι συναντήσεις με τους δύο προέδρους. Σε ό,τι αφορά την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είναι σημαντική η διαφορά που υπάρχει στην προσέγγιση μεταξύ του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας. Το Αζερβαϊτζάν έχει λιγότερες φιλοδοξίες ε, δεν επιθυμεί τόσο συμφωνία σύνδεση παρά στρατηγική εταιρική σχέση. Σε αντίθεση με την Αρμενία που τάξεται αναφανδόν υπέρ τη σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμφωνία σύνδεση. Σε ό,τι αφορά τον Αγκόνο Καραμπάχ, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την, επιστολή, την αποστολή της α, ε, ε, αντιπροσωπείας μας και μάλιστα το Αζερβαϊτζάν προσφέρθηκε να μας ε, βοηθήσει να διέρθουμε την γραμμή επαφής ενώ η Αρμενία ήταν πιο διστακτική. Πάντως ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα καταφέρουμε να περάσουμε αυτή τη γραμμή και πιστεύω ότι η Επιτροπή μας θα τα καταφέρει, επαναλαμβάνω, να διέλθει αυτή τη γραμμή επαφής και να επισκεφθεί τον Αγκόνο Καραμπάχ και από τις δύο πλευρές, και από την Αρμενία και από το Αζερμπαϊτζάν. Φυσικά υπό τους όρους και την αιγίδα του Συμπροέδρου της Ομάδας του και του Πρέσβη Λεφόρτ, τον οποίο συναντήσαμε και είχαμε μαζί του και ανταλλαγή απόψε. Θα ήθελα τώρα, εν κατακλείδη, να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Πακού και το Ιερεβάν για τη συνεργασία που είχαμε και την αμέριστη υποστήριξη των δύο αντιπροσωπιών στον Πακού από τον πρέσβη Κόμπια ε, που έδειξε υψηλό επαγγελματισμό και μεγάλη υποστήριξη και επίσης ήταν πολύ ικανοποιητικέ οι επαφές μας και στο Γερεβάν με την αντίστοιχη αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να το συζητήσουμε κιόλα. Uh, Μάλιστα. Λοιπόν. Ε, ωραία. Προτείνω να συζητήσουμε τις ε, εκθέσεις αυτές. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η κυρία Γεδανμάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ήταν εξαιρετικό το ότι αρχή αρχή ακούσαμε την ε, ενημέρωση αυτή για την κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία και νομίζω πως αυτό ξεκαθάρισε πως οι συμβιβασμοί διαφορετικών απόψεων δεν είναι πάντα κάτι το τόσο εύκολο γιατί η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν σε κάποια ζητήματα έχουν αντιδιαμετρικές απόψεις οπότε, οπότε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι εργαστήκαμε πάνω σε αυτό το θέμα. Η έκθεσή μου ε, αφορούσε το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία και χαίρομαι για το ότι τόσοι πολλοί από εσά ε, ε, είχαν ασχοληθεί με το θέμα μπορούσαμε να έχουμε και λιγότερες ε, τροπολογίε για να πω την αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει καταφέραμε να βρούμε συμβαστικέ ε, τροπολογίε. Αλλά αντιλαμβάνεται κανείς πως όταν είναι τόσε πολλέ δεν είναι και εύκολο να συμβάσουμε τις διάφορες απόψει. Αλλά με τη βοήθεια σας τα καταφέραμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους ε, ε, εισηγητές και τους σκιώδες εισηγητές και τους σκιώδες εισηγητές για την έκθεση της ε, Αρμενίας. Οπότε δεν συλλαμβάνεστε πως ε, πρέπει οι εκθέσει οι να ευθυγραμμίζονται γιατί εντάξει θα είναι διαφορετική η άποψη για τα προβλήματα αλλά μπορούμε να έχουμε και κοινέ απόψεις ε, στην ε, Ολομέλεια. Για να μην ε, έχει και το Κοινοβούλιο δύο τελείως διαφορετικές απόψεις. Το Αναγκρίνο Καραμπάχ λοιπόν ήταν το θέμα το οποίο είχε τις περισσότερες τροπολογίες και εδώ πέρα τόσο με βάση στην ομάδα του Μίνσκα η οποία εργάζεται αρκετά αργά και βεβαίω αυτό είναι πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκπροσωπείται, εκπροσωπείται η Γαλλία. Οπότε Επιθυμητό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο στην επίλυση αυτής της διαφοράς στο μέλλον. Και αυτό είναι και προς το συμφέρον της περιοχής και προς το δικό μας. Τώρα για τις λεπτομέρειες. Το, το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι το ζήτημα το οποίο προκάλεσε τις ε, περισσότερε συζητήσεις, αλλά εάν εθετηθούν οι συμβαστικές τροπολογίες 2 και 5, θα έχουν καλυφθεί ήδη πολλά ζητήματα και από ό,τι φαίνεται καταφέραμε να έχουμε μια κοινή άποψη. Παρ' αυτά θα ήθελα να τονίσω πως η συμφωνία σύνδεσης ε, δεν θα επιλύσει το πρόβλημα αυτό. Είναι δύο χωριστά ζητήματα. Η Συμφωνία Σύνδεσης είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και των χωρών αυτών και το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι διμερές. Όσον αφορά λοιπόν τα προβλήματα του Αζερβαϊτζάν, όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ε, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι και κάποιοι ε, πολιτικοί κρατούμενοι βεβαίως. Υπάρχει και το ζήτημα της ενέργειας που δεν είναι πρόβλημα βεβαίως, αλλά μας απασχολεί και η Eurovision, στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί έγιναν μέχρι και τροπολογίες ε, για μποϊκοτάζ της Eurovision. Δεν είμαι υπέρ να πω σε επιχείρημα πως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε διαφορετικούς ε, διαγωνισμούς ε, και ε, υπάρχουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, π.χ. στη Μεγάλη Βρετανία. Μόλις καταδικάστηκε η Μεγάλη Βρετανία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρόλα αυτά θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. πάντων αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γενικότερα και στις δύο αυτές εκθέσεις νομίζω υπάρχουν και θετικά και αρνητικά σχόλια με τρόπο ισορροπημένο και σας ευχαριστώ όλους. Δεν αρκεί να ευχαριστήσω μόνο έναν και δύο. Και έτσι συγκεντρωθήκαμε στα βασικά ζητήματα με τη βοήθειά σας. Βεβαίω, ε, το ζήτημα της ε, συμφωνίας ε, σύνδεσης είναι μια διαφορετική έκθεση η οποία θα μα απασχολήσει αργότερα και προς την Κομισιόν. Θα ήθελα να πω πως όταν ε, διασφαλίζει τα δικά μας συμφέροντα πρέπει να σημειώσει πως και οι δύο αυτές χώρες είναι ε, είναι Δεν ε, πρέπει να είμαστε αλαζονικοί στην εξωτερική πολιτική, να παριστάνουμε ότι ξέρουμε τα πάντα κάθε χώρα έχει διαφορετική ιστορία, εμπειρίες και μέσω της συνεργασίας μπορούμε να προοδεύσουμε, αλλά όχι να παριστάνουμε ότι ξέρουμε τα πάντα καλύτερα από όλους. Να υπενθυμίσω πως βλέπω κάποιες διαφορές μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Μεγάλης Βρετανίας παρόλα αυτά. Ε, δεν είναι όλες οι συγκρίσεις ε, σωστές. Ορίστε. Ε, ναι, ναι, έτσι. Πράγματι, έχει δίκιο ο κύριος Γκάλερ. Περνάμε τώρα στον κύριο Τάνοκ, ο οποίος ε, θα μας αναφέρει των σχεδόν Πράγματι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Υπάρχει διαφορά ε, μεταξύ των δύο χωρών. Κοιτάξτε, εμείς ε, έχουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά τα πολιτικά δικαιώματα των φυλακισμένων. Ε, κατά την άποψή μου αυτό είναι ζήτημα του Βρετανικής Βουλής και όχι ενός ε, δικαστηρίου στο Στρασβούργο. Και είμαστε και ο μεγαλύτερος επενδυτής στο Αζερβαϊτζάν, αλλά πέρα από αυτό δεν νομίζω να ωφελούν οι συγκρίσει. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη για το ότι ο συνάδελφος ε, απουσιάζει σήμερα, έπρεπε να επιστρέψει στην Πολωνία και ζητά συγγνώμη. Τον εκπροσωπώ. Οπότε ε, θα με συγχωρήσετε, δεν ξέρω τα πάντα για την Αρμενία και είμαι φίλος της χώρας αυτής. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε όλους τους γεωδησηγητές για τις 121 τροπολογίες και 10 συμβιβαστικές. Όπως ανέφερε η κυρία Γιατενμάκη, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και στις δύο εκθέσεις και ειδικά σε αυτή την έκθεση όσον αφορά την ε, συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων είναι να βρεθεί μια διατύπωση η οποία θα ε, ε, μπορέσει να ισχύσει για το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Περίεργο. Μα όταν ήμουν νέος, εμείς ε, ε, λέγαμε τα περίεργα και μυστήρια πολιτικά ζητήματα, τα λέγαμε να γκορνό Καραμπαχοειδή, το καιρό εκείνο. Αλλά αυτά ήταν, ε, αυτό ήταν απλά για να σας πω πόσο καιρό διαρκεί αυτή η σύγκρουση. Αυτό η ψηφοφορία δεν είναι αύριο νομίζω στην Επιτροπή, είναι αύριο. Οι ημερομηνίε αυτή τη στιγμή είναι οι εκλογές στις 6 Μαΐου, βουλευτικές εκλογές Αρμενίας. Και υπάρχουν διαβεβαιώσεις πως θα γίνουν με τρόπο δίκαιο, διαφανή τα Και, και θα υπάρξει και μια αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών ε, για να τις παρατηρήσει κάτι το σημαντικό για την Αρμενία. Η Αρμενία, για όσους δεν ξέρουν τη γεωγραφία τους, ε, είναι μια μικρή χώρα. Ο πληθυσμός, τον ακριβή πληθυσμό δεν τον ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέλος Συμβουλίου της Ευρώπης, ο ΑΣΕ της Ανατολικής Γειτονίας και βεβαίως ε, στο Νότιο Κάυκασο τα ζητήματα είναι και η διμερή σχέση των χωρών με τις Βρυξέλλες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστούν μεταξύ τους, ακόμα και σε στρατηγικά ζητήματα όπως η ενέργεια κτλ. Και, κατά την άποψή μου, υπάρχει ένα ε, ζήτημα που, με το οποίο συμφωνούν και οι γειτονικέ χώρες, όπως ε, η Γεωργία παραδείγματο χάρη, πως συχνά η Αρμενία μεταξύ Γεωργίας, Αζερβαϊτζάν και Τουρκίας ε, έχει βρεθεί στριμωγμένη ειδικά όσον αφορά τους ε, ενεργειακούς ε, διαδρόμους. Αν δούμε παραδείγματος χάρη τον αγωγό της BP από Μπακού, Τυφλίδα, Τσεϊχάν, είναι πάρα πολύ μεγάλη επένδυση, αλλά δεν έχει πρόσβαση η Αρμενία και βασίζεται σε ρωσικές και ιρανικές προμήθειες, συν έναν παλαιό σοβιετικό πυρηνικό αντιδραστήρα σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι ε, ρήγμα σεισμικό και τώρα υπάρχει μια δέσμευση ε, ε, περί κλεισίματος του αντιδραστήρα μέχρι το 2016. Η Αρμενία θέλει πολύ αυτή τη συμφωνία σύνδεσης και την βαθιά και σφαιρική ζώνη ελευθερίου εμπορίου και την απελευθέρωση της βίζας και συμφωνίες σε όλο αυτό το πακέτο που υπογράφουμε τώρα με τις πρώην Σοβιετικές χώρες ε, και η Ουκρανία τα ίδια ε, είχε, ε, είναι δηλαδή τα τυποποιημένα πράγματα για να έχουμε καλές εμπορικές σχέσεις με διαστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και το όλο ζήτημα επανεισδοχής και διευκόλυνσης παροχής βίζας ε, και επελευθέρωσης αυτής. Το όλο ζήτημα Αρμενίας ε, Ναγκόρνο Καραμπάχ, ε, έτσι για μένα, φιλοσοφικά, είναι το δίλημα μεταξύ της αυτοδιάθεσης ως απόλυτης αρχής και της εδαφικής ακαιρεότητας. Βεβαίως ως ρεαλιστής πολιτικός ξέρω πως καμία από αυτές τις αρχές δεν είναι απόλυτη, πρέπει να κρυθούν τα πράγματα κατά περίπτωση, λαμβάνοντα υπόψη και την ιστορία και τα διάφορα συμφέροντα και παράγοντες. Γι' αυτό νομίζω πως και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται από κοινού όταν περιγράφουμε το ζήτημα του Νεγκόρνο Καραμπάχ για να μπορέσουμε να συμβάσουμε διαφορετικές πολιτικές απόψεις και να λάβει υπόψη βεβαίω και τον αιματηρό πόλεμο που έλαβε χώρα πριν από 20 χρόνια. Εμεί στο Κοινοβούλιο συμφωνούμε σε κάτι. Η ομάδα του Μίνσκ που είναι η βασική ομάδα διαπραγμάτευσης ε, του ζητήματος αυτού ε, πρέπει να παραμείνει αυτή παρά το ότι θέλουν κάποιοι εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ και η ομάδα μου θεωρούν πως δεν πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα από την ομάδα του Μίτσελ. Να υπενθυμίσω πως η Γαλλία είναι ε, ε βασική χώρα εκεί πέρα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπε η κυρία Γιατερμάκη για την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτραπεί και στις δύο εκθέσεις να χρησιμοποιηθεί η ίδια ορολογία, αλλιώς ε, θα υπάρχει ασυνέπεια στο έργο της Επιτροπής και οπωσδήποτε θα προκαλώσει ατέρμονες συζητήσει στον τύπο Αρμενία και Αζερβαϊτζάν για το τι είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά έχουμε 10 συμβιβαστικέ τροπολογίε, υπάρχουν 121 βεβαίω από αυτές. Φαντάζεστε πως τα περισσότερες είναι απλές, πλην του ζητήματο του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ε, νομίζω πως θα δείτε το τελικό αποτέλεσμα την υπαριθμών 6 βασική συμβαστική τροπολογία που προσπαθεί να συμπεριλάβει τα πάντα. Μία ενιαία διατύπωση, αλλά και εδώ πέρα υπάρχει έτοιμα για χωριστία σε τμήματα. Αλλά να πω πως ε, σύμφωνα με την άποψη της ομάδας μας ε, και του ΣΥΚΤΟΥ είναι ένα πακέτο. Εάν διαλύσουμε την συμβαστική τροπολογία είναι δύσκολο να ε, συμφωνήσουμε μετά όλες οι ομάδες. Πρέπει να μείνουμε σε αυτή τη εντύπωση. Αυτά είχα να πω. Θα σημειώσω τα σχολεία των συναδέλφων και σχεδόν εισηγητών για να τα μεταφράσω στον συνάδελφο. Ευχαριστώ. Είμαι Μακοβέη. Thank you. Um, never be let, you never stop on Mr. Preda. I'd like to say a few words on Azerbaijan. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για το Αζερβαϊτζάν, όπου είμαι σκιώδης εισηγήτρια και συμμετείχα σε αυτήν την επίσκεψη αποστολή στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Καταρχήν είναι σαφές για όλους μας ότι η εταιρική μας σχέση με το Αζερβαϊτζάν θα πρέπει να βασίζεται σε κοινέ αξίες, δηλαδή σεβασμός δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα. Το Αζερβαϊτζάν κατέστησε σαφή την πρόθεσή του να σεβαστεί όλες αυτές τις αξίες και να εκδημοκρατιστεί. Όμως υπάρχουν πολλά ακόμα προβλήματα και αναφέρονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χώρα αυτή είναι ανεξάρτητη μόνο εδώ και 20 χρόνια. Ωστόσο, περιμένουμε μεγαλύτερες προσπάθειες και αυτά τα θέματα να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα, σε σχέση με την ε, συμφωνία σύνδεσης, την οποία διαπραγματεύεται η Κομισιόν και που όπως ακούσαμε από τον κύριο Κοβατσέφ, το Αζερβαϊτζάν δεν είναι και πολύ πρόθυμο να την φτιάξει, δεν ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Εγώ δεν είμαι βεβαία. Χρειαζόμαστε νομική βάση για τη συνεργασία μας. Θα μπορούσε αυτή να είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση, αλλά δεν θα έλεγα ότι το Αζερβαϊτζάν δεν ενδιαφέρεται για μια συμφωνία σύνδεσης η ιδέα είναι ότι αν θέλουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι μπορούμε σε μια τέτοια συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά την διευκόλυνση θεωρήσεων ε, και τη σχετική συμφωνία, ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις 7 Μαρτίου. Αυτό είναι κάτι το νέο, λοιπόν. Και Βασικά θα διευρύνει τη συζήτησή μας και τον διάλογο περί κινητικότητας για τη συνεργασία για την ενέργεια. Το Αζερβαϊτζάν, μάλλον εταιρική σχέση ε, Αζερβαϊτζάν-Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει. Το Αζερβαϊτζάν ήταν ασθενό εταίρο και εξασφάλισε τη διαφοροποίηση των, των εφοδιασμού ενέργεια ε, στην, ε, στην Ευρώπη. Κυρία Μακοβέη, μπορείτε να εστιάσετε την προσοχή σα στι τροπολογίε. Ναι. Ναι να αναφερθώ στι ε, τροπολογίε για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ε, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η αποστρατιωτικοποίηση, ε, η απόσυρση των αρμενικών στρατικών δυνάμεων από τον Αγκόρνο Καραμπάχα και ε, από την περιοχή θα είναι ε, πολύ σημαντική. Επίσης, πρόληψη περιστατικών και μηχανισμός ε, πρόληψης της παραβίασης της ανακοχής, η επιστροφή των προσφύγων στις αιστείες τους και η πολυεθνική δύναμη επιχείρηση μάλλον διατήρηση της ειρήνης για να τα επιβλέπει όλα αυτά ώστε να γίνουν ομαλά. Τις τροπολογίες θέλω να πω ότι κάτι λείπει για παράδειγμα, η απόσυρση των αρμενικών δυνάμεων ε, φέρουν την απόσυρση των δυνάμεων αυτών μόνο γύρω από τον Αγκόρνο Καραμπάχ και όχι από το ίδιο τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Νομίζω πως είναι λάθος αυτό. Τεχνικής φύσης. Και επιμένω για αυτά που συμφωνήσαμε χτες στην τελευταία συνεδρίαση για αυτή την ε, επιχείρηση, πολυεθνική επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης, της την ειρηνευτική αυτή επιχείρηση. Δεν νομίζω πως θα πρέπει να επιμείνουμε τώρα για δημοψήφισμα ε, το οποίο θα καθορίσει την ε, θέση και θα παρέχει την νομική βάση για τη χώρα αυτή. Αν είδα καλά τις συμβαστικές τροπολογίες υπάρχουν εκεί πέρα κάποια σημεία των ε, αρχών του Μίνσκ και της δήλωσης αυτής νομίζω. Κύριο Σαλάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα στραφώ άμεσα στις ε, τροπολογίε, γιατί νομίζω πω η γενική συζήτηση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Και να πω μόνο μία σκέψη. Πιστεύω πως είναι μια πολύ καλή δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ετούτε εδώ. Έχουμε ολοκληρώσει πολύ δύσκολες αλλά δίκαιες διαπραγματεύσει ανάμεσα στις ομάδες και έχουμε φτάσει σε μια κοινή θέση που αφορά το θέμα της συμφωνίας με το Αζερβαϊτζάν και την, Αρ... την Αρμενία. Το γεγονός ότι αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε το ίδιο κείμενο είναι επίσης πολύ σημαντικό για τα διάφορα θέματα κλειδιά. Έχουμε ξεκάθαρη θέση του Κοινοβουλίου που είναι ε, αυτό πολύ καλή συμβολή ώστε να ε, γυρίσουμε σελίδα πια, στο, ειδικά για το θέμα του Νακόρνου Καραμπάχ, για αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα, ε, δηλαδή την ε, ανεφοδιασμό σε ενέργεια και τον Νακόρνου Καραμπάχ, έχουμε δύο τροπολογίες ε, πολύ σωστές. Ο συνάδελφος του ΕΛΚ ήδη περιέγραψε τα πιο σημαντικά θέματα που είναι πολύ χρήσιμο αυτό γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα. Και λεπτομερή όσον αφορά το θέμα. Το θέμα της ε, διαφοροποίησης της, ε, του ανεφοδιασμού ενέργειας πιστεύω πως η συμβιβαστική τροπολογία παριθμών 6 ε, αναπτύσσει μια ποσοστή και λογική θέση. Και άρα αυτό θα γίνει δεκτό στην περιοχή ως μια σοβαρή συμβολή του Κοινοβουλίου για την ειρηνική λύση των προβλημάτων της περιοχής. Ελπίζω λοιπόν και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια ελπίζω πως δεν θα ε, ακυρώσει όλη την προηγούμενη δουλειά που έχουμε κάνει. Thank you. I Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και τους δύο για το έργο τους. Δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα, γιατί πήγαμε και στις δύο χώρες και εξαιτία της σύγκρουσης στον Αγκόνο Καραμπάχ υπάρχει κάτι που ισχύει και για τις δύο χώρες. Και θα πρέπει να τα εντάξουμε στα ψηφίσματα με τις συμβαστικές λύσεις. Νομίζω ότι το συνολικό πακέτο είναι ικανοποιητικό. Να ξεκινήσω με τις συμβαστικές τροπολογίες. Συμφωνώ με την τροπολογία 2 για το Αζερμπαϊτζάν και την 6 για την Αρμενία. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Έχω όμως ακόμη ένα πρόβλημα και περιμένω τις απόψεις των συναδέλφων. Έχω πρόβλημα με το τελευταίο εδάφιο Εκεί μιλούμε για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος μετά την επιστροφή των προσφύγων. Θα ζητήσω ψηφοφορία κατά τμήματα και ξεχωριστή ψηφοφορία για το συγκεκριμένο εδάφιο. Γιατί λέμε προκειμένου να δημιουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις για την ε, έκφραση ελεύθερης ε, βούλης του, λα του λαού σε ό,τι αφορά την θέση του Ναγκόνο Καραμπάχ. Συμφωνώ με την ελεύθερη θέληση, έκφραση ελεύθερης βούλησης κτλ. Αλλά όταν ε, συγκρίνουμε με άλλες περιπτώσεις όπου είχαμε σύγκρουση, πόλεμο, ε, κατοχή και μετά δημοψήφισμα, το θέμα είναι ποιος ε, αποφασίζει στο δημοψήφισμα. Οι, αυτοί που διαμένουν τώρα, αυτοί που έχουν επιστρέψει, τα παιδιά των ε, προσφύγων που έφυγαν και ίσως γυρίσουν. Ποιος θα ψηφίσει, ποιος θα λάβει μέρος σε αυτό το δημοψήφισμα. Και έχουμε προβλήματα όπως η Δυτική Σαχάρα που έχουν μείνει ανεπίλητα. Να ζητήσουμε δηλαδή κάτι, ένα δημοψήφισμα που ξέρουμε ότι θα είναι προβληματικό, δεν ξέρω. Γι' αυτό θα ζητήσω ξεχωριστή ψηφοφορία του σημείου αυτού συνήθι μια συμφωνία, αλλά εγώ δεν συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις. Κάποιες ομάδες μόνο συμφώνησαν. Ε, εγώ δεν έδωσα τη γνώμη μου. Έχω ένα πρόβλημα με τη διατύπωση και θα ζητήσω ξεχωριστή ψηφοφορία. Για τους λόγους που σας είπα, δεν είμαι κατά της διεξαγωγής δημοψηφίσματος γενικώ. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση οι λεπτομέρειες είναι πολύ δύσκολες και θα οδηγήσουν σε αναβολή των αποφάσεων και των πολιτικών και των άλλων. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Τώρα, για κάποιες άλλες τροπολογίες που κατέθεσα με συναδέλφους και που δεν καλύφθηκαν από τις συμβαστικές τροπολογίες. Και θα ζητήσω την υποστήριξή σας. Η μία από αυτές είναι πολύ σημαντική, αφορά το Αζερμπαϊτζάν και παροτρύνει τις ε, αρχές του Αζερμπαϊτζάν να εκτελέσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόσφατα ε, οι δικηγόροι μίλησαν για την υπόθεση δύο αδερφών που είναι φυλακισμένοι εδώ και χρόνια και το 2010 και 2011 ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, κήρυξε ένοχο το Αζερβαϊτζάν για τη μη διεξαγωγή δίκαιη ε, δίκη και ζήτησε απελευθέρωση των δύο αδελφών και αποζημίωσή του. Τίποτα δεν έχει συμβεί, δεν έχει εκτελεστεί αυτή η απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι στη φυλακή. Γι' αυτό παρακαλώ να εγκρίνετε τη σχετική μου τροπολογία. Κάτι άλλο πάλι για το Αζερβαϊτζάν. Το θέμα του ειδικού εισηγητού της κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για ε, τους πολιτικούς κρατουμένους. Ζήτησε πρόσβαση στις φυλακές, κάτι που του απαγορεύθηκε από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν. Αυτό επισημένω στην τροπολογία μου, παρακαλώ να την υπερψηφίσετε. Κατέθεσα και τροπολογίες που είναι κοινέ, ισχύουν και για το Αζερμπαϊτζάν και για την Αρμενία. Μία από αυτές ε, είναι η παριθμόν 72 για το Αζερμπαϊτζάν, ζητά το σταμάτημα της, ε, ε, του εξοπλισμού, του στρατιωτικού εξοπλισμού και ζητά από τις ε, ευρωπαϊκές χώρες να μην εξάγουν όπλα. Γιατί η αύξηση του στρατιωτικού προϋπολογισμού και των δύο χωρών δημιουργεί ανησυχίες για την καθυστέρηση στην, στο διακανονισμό των, της εκκρεμού σύγκρουσης. Γι' αυτό ζητώ από τις χώρες να σταματήσουν να εφοδιάζουν τις χώρες αυτές με όπλα. Δεν νομίζω ότι είναι δόκιμη αυτή η συνέχιση της εξαγωγής όπλων προς τις δύο χώρες. Ένα άλλο θέμα. Το Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο. Θα ήθελα να υπερψηφίσετε αυτή την τροπολογία, γιατί τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν γνωρίζουν σύνορα. Και νομίζω ότι για αυτό το ζήτημα απαιτείται πλήρη συνεργασία. Και τελευταίο σχόλιο, παρακαλώ ψηφίστε την τροπολογία μου για την Ερμηνεία και για το κλείσιμο του πυρηνικού εργοστασίου του Μετζαμόρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τα καλά σας αγγλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας αγγλικά να υπενθυμίσω κάτι. Εδώ πέρα μιλάμε για τις βασικές αρχές της ομάδας του Μίνσκ και μετά διαγράφουμε αυτές που δεν μας αρέσουν. Ε, πρέπει να σας πω κάτι. Σπάνια στην πολιτική μου ζωή μου έχει ασκηθεί τόσο λόμπινγκ όσο από αυτές τις δύο πλευρές εδώ πέρα δεν είναι σωστό, ανεξαρτήτως από ποιον προέρχεται. Ο καθένας θέλει να σβήσει μια φράση εδώ πέρα. Λέει, οι αρχές του Μίνσκ ε, θα γίνουν έτσι μη ισορροπημένες για τη μία ή την άλλη πλευρά. δεν έχει ξεκαθαριστεί το πώς θα φύγουν τα αρμενικά στρατεύματα από τις κατεχόμενες περιοχές, αλλά είναι μέρος των αρχών. Ας ε, γράψουμε λοιπόν όλες τις αρχές και να μην αναθεωρήσουμε εμεί εδώ πέρα τις αρχές του Μίνσκ ή προτείνω να βάλουμε μια τελεία μετά τη σύγκρουση του Νακόρνο Καραμπάχ, τελεία και να σβήσουμε όλο το υπόλοιπο κείμενο. Έτσι για να τελειώσουν οι καυγάδες. Δεν θα λύσουμε εδώ πέρα τη σύγκρουση αυτή. με το να βάζουμε φράσεις ε, και να αναθεωρούμε τις αρχές του Μίνσκ. Ε, δηλαδή, λάβετε το υπόψη. Ναι, αν θέλουμε να συνεισφέρουμε, πρέπει να, να γνωρίσουμε τα πάντα. Όλες τις αρχές αυτές. Όλες τις βασικές αρχές της ομάδας του Μίνσκ. Και, παρακαλώ, προσέξτε το αυτό. Αν μας βίνουμε τα κομμάτια που δεν μας αρέσουν, δεν, δεν έχει νόημα. Οπότε να αφήστε τα όλα όπως είναι μέσα ή να τα διαγράψουμε όλα. Και να μιλήσουμε γενικώ για τις αρχές. Αλλά όχι να σβήσουμε τη λέξη που δεν αρέσει τον καθένα για να έχει κάποιο λίγο πιο πολύ δίκιο. Ε, γιατί μετά δεν θα είναι αποδεκτά αυτά που γράφουμε. Αναφέρεται Κοιτάξτε, αυτό που λέει η ελεύθερη έκφραση για το τελικό καθεστώς είναι μέρος των αρχών, τις οποίες έχουμε αναγνωρίσει όλοι. Το πώς θα εφαρμοστούν μετά είναι άλλη ιστορία. Αλλά να διαγράψουμε τις αρχές δεν μου φαίνεται. Δεν είναι σωστό και δεν κάνουμε και τίποτα έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Ντόγκης τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές. Πιστεύω πως έγινε καλή δουλειά για τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Δεν ε, χρειάζεται να επαναλάβω τις παρατηρήσεις ε, των συναδέλφων για να μην ε, χρονοτριβήσω, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ένα σημείο. Από τις δύο πλευρές υπάρχουν έντονο αίτημα και από την Αρμενία και από το Αζερμπαϊτζάν για διαπραγματεύσεις όσον αφορά το Αζερβαϊτζάν για στρατηγική συνεργασία και όσον αφορά την Αρμενία για μια πραγματική σύνδεση. Θέλω να θυμίσω πως υπάρχει και ένα ανοιχτό κεφάλαιο στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, το οποίο μπορεί από την δήλωση της Πράγας. Αυτό σημαίνει μάλλον ενδιαφέρονται και, και το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία. Στην συμβαστική 6 υπάρχει ένα σχετικό σημείο και όπου λέει ότι οι διαπραγματεύσει θα πρέπει να είναι δεσμευτικέ, να συνδέονται με πιστευτές ε, δεσμεύσεις και ουσιαστικές πρόοδους. Αυτή η παρατήρηση είναι πολύ σημαντική γιατί περνά, ξεπερνά μια δήλωση αρχής. Ε, αν έμενε έτσι όπως ε, ήταν πριν, εντάξει, θα ήταν πιο αόριστο. Όμως εδώ πρόκειται για μια συγκεκριμένη δέσμευση με πολιτικό χαρακτήρα και που το ζητά η, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μπορεί να προβεί σε ε, πολιτικές δεσμεύσεις και να ζητήσει πράγματα. Από την άποψη όμως του θέματος που έθεσε ο Τάνοκα που λέει και αναφέρεται στην αυτοδιάθεση και στην εδαφική κυριότητα Αυτή είναι παλιά συζήτηση, όμως υπάρχει ένα σημαντικό ε, θέμα εδώ. Ε, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνουν διαπραγματεύσεις με βάση μια κατάσταση παρανομίας. <coughs> Ανομίας. Γιατί η διαβίες κατοχή δαφών είναι παράνομη. Και για τον ΟΙΕ και για διεθνώ, σε πάση περιπτώσει. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες βασικές, βασικοί όροι που θα πρέπει να τους σεβαστούν. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι έτσι πως Έχουμε πει επανειλημμένα για την Γεωργία ότι θα πρέπει να υπάρξει απόσυρση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ζητήσουμε στον Αγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο είναι υποκατοχή, να πούμε ότι προϋπόθεση θα, για τις διαπραγματεύσεις θα είναι η απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων. Συμφωνώ με τη Λούνατσεκ για ένα δημοψήφισμα ένα δημοψήφισμα μπορεί να αλλάξει αν δεν βρεθούν οι κατάλληλοι, αν δεν ισχύουν μάλλον οι κατάλληλοι όρια. Αν ένα δημοψήφισμα γίνει συγκεκριμένη μέρα και όχι κάποια άλλη και αφήσουμε να περάσει πολύ καιρό, είναι σαφές ότι οι προποθέσει διαφάνειας αυτού του δημοψηφίσματος μπορεί να αλλάξουν. Στην Δυτική Σαχάρα έχουμε ένα απτό παράδειγμα για τα όσα λέω. Αυτά θα ήθελα να πω. Έχω κι άλλα να πω, αλλά θέλω να σεβαστώ τον χρόνο που μας έδωσε ο Πρόεδρος Μπρόκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να πω τρεις παρατηρήσεις να κάνω για την αποστολή Κοιτάξτε, υπάρχει στασιμότητα στον Αγκόνο και θα λυθεί υπόψη ως πακέτο. Δεν υπάρχει ένα κομμάτι μόνο. Οπότε έχει δίκιο εδώ πέρα ο Θα αναφερθούν όλες οι αρχές του Μίνσκ και καμία. Δεν έχει νόημα να επιλέγουμε. Ή όλα ή τίποτα λοιπόν. Δύο παρατηρήσεις λοιπόν. Ο πρόεδρος Αλίγεφ δεν είπε πως η Γαλλία πρέπει να την από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε πως είναι εκεί πέρα ο Μετβέντεφ και όχι ο Ομπάμα ή ο Σαρκοζή, παρά μόνο οι πρέσβεις. Και ήταν κάπως μονομερή τα πράγματα. Αλλά δεν είπε να αντικατασταθεί η Γαλλία. Βεβαίω, όπω ε, λέει η συνθήκη τη Λισαβόνα, η Γαλλία πρέπει να εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Από την άλλη, δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν εδώ πέρα εντελώς, γιατί ε, ε, εμείς είπαμε πως θα έπρεπε να διάσει μια επαρχία από τον αρμενικό στρατό και λέτε πως δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση ο Αρμένιος πρόεδρος. Ήταν ξεκάθαρη απάντηση και είπε όχι. Γιατί είπε πως αν ε, φύγει από μία επαρχία γιατί να μην ε, φύγουν και από τις άλλες. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Είναι μία σκληρή γραμμή και μία λύση πακέτο ή τίποτα θα δοθεί. Ο Δέλμαρ Μπρόκ ε, έχει δίκιο, πρέπει να κινηθούμε στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει, δεν έχει να κερδίσει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κάποιος ο οποίος θα παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο εδώ πέρα. Δεύτερη παρατήρηση συμφωνία σύνδεσης. Ακούστηκε πως έχει προχωρήσει πολύ η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν δεν θέλει καν συμφωνία σύνδεσης. Ο Υπουργός, δε, ο κύριος ε, Χαζημός, ε, μας είπε επιλέξει, μου, μου φέρατε κάτι από τις Βρυξέλλες που δεν μου χρησιμεύει τίποτα. Δεν το θέλω αυτό. Εντάξει, στρατηγικό εταίρο για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, εντάξει. Αλλά αυτά τα πράγματα τώρα που μου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ πέρα, αξίε και αρχέ και τέτοια, τι να τα κάνω. Οπότε οι τροπολογίε μα έχουν εδώ πέρα έχουν ένα πρόβλημα. Γιατί η συμφωνία σύνδεση θέλουμε να συνδεθεί με ειρηνική λύση, Αλλιώ δεν θα υπάρξει ε, τέτοια συμφωνία. Μα όταν ε, θα χρειαστεί σε ένα χρόνο το πολύ να δούμε αν θα μπλοκάρουμε τη συμφωνία σύνδεση γιατί δεν θα έχουν οπωσδήποτε ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει. θα πρέπει να σκεφτούμε θέλουμε να μπλοκάρουμε όντω τη συμφωνία ε, λόγω τη καστέρησης με το Αζερβαϊτζάν ε, γιατί το Αζερβαϊτζάν δεν θέλει καν τρίτη παρατήρηση για την πολιτική κατάσταση πράγματι η κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν είναι ε, επισφαλής. Ε, εμείς θεωρούμε πως δεν θα πρέπει να υπάρξει μποϊκοτάς της ε, Eurovision. Ε, πρέπει να την εγκαταλευτούμε. Υπάρχουν διάφορες ομάδες που λένε τραγουδώντας για τη δημοκρατία και τέτοια. Είναι μια κάποια πρόοδος μπορεί να σημειωθεί σε ζητήματα ελευθερίας γνώμης. Ε, στον Αζερβαϊτζάν μιλάνε για καμπάνια κατά της χώρας. Δεν συμβαίνει αυτό, αλλά δεν είναι και σωστό να μποϊκοτάρουμε το διαγωνισμό. Κοιτάξτε, θα περιοριστούμε σε δύο λεπτά να ομιλητή, αλλιώς δεν θα τελειώσουμε. Είναι πάρα πολλοί ομιλητές. Ο κύριος Κυρίλοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια και είμαι ο πρώτος με τον περιορισμένο χρόνο ο πρώτος ομιλητής. ήθελα να πω ότι μετά την έκθεση για την ανάγκη νέας ε, ευρωπαϊκής στρατηγικής στο Νότιο, στο Νότιο Κάφκασο που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία συμβάλλουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα πιο ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Νότιο Κάφκασο θα... και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έκκλησης και με την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι πιο δραστήρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπουμε και πολιτικά μηνύματα και στις ανακοινώσεις αλλά και από τις τελευταίες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, οι δύο εκθέσεις που εξετάζουμε σήμερα επίσης θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή και με την επίσκεψη της αντιπροσωπής της ΑΦΕΤ στην περιοχή νομίζω ότι επηρεάσαμε ε, τις εξελίξεις ε, για μια πιο ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, περιοχή. Χρειαζόμαστε τώρα υποστήριξη των συμβαστικών τροπολογιών προκειμένου να φανούμε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Είναι σημαντικό να ε, συγκεντρώσουμε μεγάλη πλειοψηφία για τι συμβαστικέ λύσεις. Συμφωνώ και εγώ ότι μερικά ζητήματα ίσω είναι συζητήσιμα περαιτέρω και δεν ε, αναφέρθηκα στην έκθεση. Στην Αρμενία ακούσαμε πολλές φορές το επιχείρημα και το παράδειγμα του Κωσυφοπεδίου. Θα πρέπει να αποτρέψουμε εδώ τέτοιες, τέτοιους παραλληλισμούς. Θα πρέπει να συμβάλλουμε σε μια πιο ενεργό παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και να ενθαρρύνουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Φυσικά επενώντας και τις δραστηριότητες της ομάδας του Μίνσκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα είμαι λακωνική. Δεν νομίζω ότι ε, έχει νόημα να συζητούμε την ε, Eurovision γιατί υπάρχει πολιτική υποστήριξη για τις ευρωπαϊκές ε, αξίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διοργάνωση του δημοψηφίσματος, δεν έχει νόημα να εξετάζουμε στην έκθεση αυτή τη σκοπιμότητα του δημοψηφίσματος. Το δημοψήφισμα είναι μια πολιτική λύση που έχουν δεχτεί και οι δύο πλευρές και θα ε, βρεθεί κατάλληλη στιγμή για τη διεξαγωγή του. Αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, δεν είναι όριμη η κατάσταση για ένα δημοψήφισμα, προκειμένου να εφαρμοστεί η λαϊκή βούληση. Κινδυνεύουμε να επιδεινώσουμε τα πράγματα, αντί να βρούμε μια καλή λύση. Θα πρέπει να τηρηθούν ε, ε, αυστηρά οι αρχές της ομάδας του ΜΙΣ και στις εκθέσεις. Βέβαια η ομάδα του Μίσκ μάλλον χορεύει παρά ε, σημειώνει βήματα προέδρου, αλλά νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε στην ανέβρεση λύση. Επίση πρέπει να ξεκινήσουμε από μια ιστορική πραγματικότητα την ανάγκη απόσυρσης των στρατευμάτων από την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Γιατί αν δεν αποχωρήσουν ε, τα στρατεύματα, δεν θα δημιουργηθεί πρόσφορα έδαφος για την ανέβρεση ειρηνικής λύσης. Είναι σημαντικό λοιπόν να το τονίσουμε αυτό και για τις τρεις χώρες. Τώρα, κατά πόσο είναι σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Νότιο Κάφκασο, τι να σας πω, πολλά από τα αιτήματά μας ε, παραβλέφθηκαν. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις προτεραιότητές μας και να υιοθετήσουμε και μια ελαστική προσέγγιση. Πιστεύω πάντως ότι ο Κάφκασος ε, μας δίνει μια ευκαιρία στην πολιτική γειτονία και θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τις χώρες της περιοχής. Ευχαριστώ. Πολλά ακούσαμε για το θέμα αυτό ήδη. Και θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου προς τους ηγητές και τους σκιώδεις ηγητές για τις ε, σοβαρές προσπάθειες που κατέβαλαν μέσω των συμβαστικών τροπολογιών να συσπυρώσουν ε, τους ευρωβουλευτές προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι πολύ δραστήριο και να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής και όχι απλώς να μιλά για την ευρωπαϊκή προοπτική των δύο χωρών. Πάντως, το βασικό πρόβλημα και των δύο χωρών είναι τον Αγκόνο Καραμπάχ. Και συνεχίζω τις σκέψεις του κυρίου Προβέρα θα πρέπει να σεβαστούμε τα μέχρι τώρα επιτέγματα της ομάδας του Μίνσκ. Αλλά κολλησιέργησε κάπως η ομάδα του Μίνσκ. Νομίζω ότι ήταν υπερβολική αυτή η καθυστέρηση. Και στο μεταξύ η κατάσταση έχει αλλάξει επί τόπου. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εθνοτική κατάσταση στον Αγκόνο Καραμπάχ. Οπότε, αν θέλουμε κάπως να βελτιώσουμε τις συμβεστικές τροπολογίες, καλό θα ήταν να αναφερθεί η απόσυρση ε, των αρμενικών στρατευμάτων από το σύνολο του Ναγκόρνο Καραμπάχ και όχι από τις ε, μεθόριες περιοχές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης, να ε, κάνουμε μνήμα των αρχών του διεθνούς δικαίου. Η κατοχή είναι απαράδεκτη, ιδιαίτερα ε, πολλά τα μάλλον που υποστηρίζεται από την παρουσία και ρωσικών στρατευμάτων στην Αρμενία. Κάτι που μετατρέπει την Αρμενία σε δορυφόρο της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Βάιντερ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους ε, εισηγητές, ε, τους κοιόδης εισηγητές. Η δουλειά, της είναι, η δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολες και οι χώρες. Εγώ επισκέφτηκα πρόσφατα την Αρμενία μετά από πρόσκληση της Euronest ε, κυρίως για κοινωνικά ζητήματα αλλά και εκεί πέρα ε, προέκυψε το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ και πρέπει να το λύσουμε ή να έρθουμε πιο κοντά σε μια λύση. Πρέπει να τεθεί το ερώτημα, θέλουμε η κατάσταση να μείνει ως έχει ή ε, να οδηγηθούμε σε μια λύση. Θεωρώ πως πρέπει να αναζητήσουμε μια λύση που θα αποτελέσει βάση για καλή συνεργασία μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Θα πρέπει επίσης να φύγουν τα στρατεύματα από ολόκληρη την περιοχή και να αντικατασταθούν από διεθνή ειρηνευτικά στρατεύματα και μέσα οικοδόμησης εμπιστοσύνη. κύριος Τσέκ και ο κύριος Προβέρα πρότειναν ένα δημοψήφισμα σε μια περιοχή η οποία είναι κατεχόμενη. Αυτό είναι επικίνδυνο και είχαμε εμπειρία στη χώρα μου. Μετά την κατοχή η ε, Λετονοί στα ανατολικά της χώρας είναι μόνο 15% και οι Ρωσόφωνοι 85%. Τι θα γίνει εκεί εάν γίνει ε, δημοψήφισμα. Είναι επικίνδυνο αυτό. Είναι νωρί για δημοψήφισμα στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Η δε δουλειά της ομάδας του Μίνσκ είναι ασύμετρη. Ή μάλλον ασύμετρη είναι εκπροσώπηση. Ο, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό θα έλεγα πως Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ομάδα του Μίνσκ. Υποθέτω, πως λέτε, πως δεν αναγνωρίζετε τα αποτελέσματα της ομάδας του Μίνσκ. Ε, είπα αυτό το οποίο είπα, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω πώς το ακούσατε. Δεν είναι γραμμένο σε πέτρα. Είπα πως δεν είναι όλες οι αρχές ίσως πολύ χρήσιμε σε αυτή την κατάσταση. Ναι, ναι, καλά άκουσα. Λοιπόν, κύριε Λαντσμπέργκης. Ε, thank you, President. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση για τη συμφωνία σύνδεσης ε, με το Αζερβαϊτζάν ως πακέτο σημαίνει σημαντική πρόοδο προς την πραγματικότητα και προς τη ε, αναγκαία βήματα για την εξέβρεση μιας λύσης, όχι μόνο για τον αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά και γειτονικές, ε, ε, γειτονικά κατεχόμενα εδάφη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υπάρχουν ακόμα σοβαρότερο πρόβλημα για την Αρμενία ειδικότερα. Αλλά αν αναφέρουμε την ομάδα Μίνσκ, στις συζητήσεις που γίνονται εδώ, εγώ θα έλεγα ότι να επενούμε την ομάδα του Μίνσκ δεν αρκεί. Θα πρέπει να δούμε και την ανεπάρκεια του. Αν βασιστούμε μόνο στο Μίνσκ, δεν θα πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες για την επίλυση της ε, σύγκρουσης εκεί, γιατί πρόκειται για μια ομάδα που δεν επιθυμεί την λύση. Έχουν εκεί δικά τους συμφέροντα, κυρίως την πώληση όπλων. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα επιπλέον διεθνές σώμα ειρηνευτικό. στην συμβιβαστική 5 ιδιαίτερο, που λέει επιμένουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει ισχυρότερο ρόλο. Συμφωνώ, αλλά εδώ ένα στοιχείο θα μπορούσε να διορθωθεί. Το πώς δηλαδή θα παίξει αυτό το σημαντικότερο ρόλο, υποστηρίζοντας την εφαρμογή αλλά και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες αναβαλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνη, για το πώς δηλαδή θα μπορέσουν να συμβιώσουν οι κοινότητε του Αζερβαϊτζάν και τη Αρμενία. Και πρέπει να διευκρινίσουμε τι είναι η κοινότητα των ε, ε, Αζερβαϊζανών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εκδιωχθεί, ναι, αυτοί είναι και θα πρέπει να το πούμε. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς λοιπόν για το τι Μιλάμε ακόμα για ένα θέμα για την ελεύθερη πρόσβαση της Ένωσης να διασχίζει αυτά τα εδάφη. Αυτό είναι πολύ έντονο και πρέπει να τους πιέσουμε. Εδώ δεν πρέπει να πιέσουμε το Αζερβαϊτζάν, αλλά την Αρμενία. Η Αρμενία μπλοκάρει. Σας παρακαλώ να την ολοκληρώσετε. Αν η Αρμενία μπλοκάρει την ε, πρόσβαση, θα πρέπει να το πούμε. Παρακαλώ να μείνετε στο χρόνο σας, γιατί την επόμενη φορά θα σας κόψω, γιατί δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε όλους όσους ζήτησαν το λόγο. Okay. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να βαθύνουμε τις σχέσεις μας και με τις δύο χώρες. Επίσης, θα ήθελα η διαδικασία αυτή να χρησιμοποιηθεί και για τις ε, σχέσεις καλή γειτονία και για τη μεταλαμπάδευση του ευρωπαϊκού πνεύματος. Ε, νομίζω ότι οι συμβαστικές τροπολογίες βελτιώνουν την έκθεση, δικαστούν πιο ισορροπημένοι και είμαι υπέρ. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα, συμφωνώ, Πρόεδρε, μαζί σας, ότι καλό θα ήταν να εξηγήσουμε σαφέστερα τους στόχους και τις αρχές αντί να μιλάμε μόνο για τους στόχους που μπορεί να διαφέρουν και κάποιες ομάδες πίεσης. Θα πρέπει η έκθεση αυτή να ανταποκρίνεται στη δική μας βούληση, όχι τις ιδέες κάποιων άλλων. Και να δημιουργήσουμε και ένα πρόσφορο κλίμα για την ανέβρεση λύσεων. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία με πιο ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Uh, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου που εργάστηκαν για τι συμβιβαστικέ τροπολογίε και ειδικά τη συμβιβαστική για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε ένα συνεπέ και σταθερό μήνυμα για αυτή την σύγκρουση και την επίλυση τη. Είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε για πρόσβαση της Ένωσης στον Αγκόρνο Καραμπάχ και για πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Αγκόρνο Καραμπάχ. να πω ότι έγινε μια συνόδος κεκλεισμένων των θυρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στο Αζερβαϊτζάν όσο και στην Αρμενία χτες στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εντυπωσιάστηκα με τις πληροφορίες που πήραμε και θα πρέπει να πω ότι οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να γίνει ο διαγωνισμός της Eurovision ε, γιατί είναι μια ευκαιρία ώστε να δοθεί πλήρης μας προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊσάν όπου η κατάσταση είναι χειρότερη και όπου η προθυμία να μιλήσουν και για να ξεκινήσουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι λιγότερο εμφανής από ό,τι στην Αρμενία. Επίσης, να πω ότι υπάρχει το θέμα των αδελφών Αλιέχ που ανέφερε η κυρία Λούνατζεκ. Καντίτζα Ισμαήλ είναι μια άλλη περίπτωση και εσείς την αναφέρετε κύριε Μπρόκ που είναι μια ναι, δημοσιογράφος που είναι γνωστή για τις ερευνητικές, ε, τα ερευνητικά του ρεπορτάζ και τώρα ε, εκβιάζεται. Ε, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και ελπίζω πως θα γίνει λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία γιατί φυσικά το Κοινοβούλιο δεν θα επιτρέψει ελπίζω οικονομικά προβλήματα, να καταπνίξουν αυτό το λαό που αγωνίζεται για την επικράτηση του κράτους δικαίου και για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Κυρία Ιμπρισάτζιτς. ευχαριστώ. Why we in... Θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση. Γιατί την τελευταία εκδοχή της ε, Συμβαστικής Τροπολογίας 6 αναφέρθηκε η ε, απόσυρση των αρμενικών στρατευμάτων από, το, από τις περιοχές που περιστοιχίζουν τον αγώνο Καραμπάχ. Αυτό είναι μια καινούργια διατύπωση. Είχαμε αντίστοιχη περίπτωση αλλού και συμφωνήσαμε ότι για, και για τις τρεις χώρες, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία, θα ζητήσουμε, για, θα ζητήσουμε την απόσυρση των στρατευμάτων από όλα τα κατεχόμενα εδάφη. Τώρα, αντί να λέμε από όλα τα κατεχόμενα εδάφη, λέμε από τα γύρω του Ναγκόνο Καραμπάχ εδάφη. Surrounding occupied regions. Δηλαδή, να ζητήσουμε από την Αρμενία πως ήρθε τα στρατεύματά της από τις γύρω κατεχόμενες περιοχές του Ναγκόνο Καραμπάχ, δηλαδή ε, δεχόμαστε να παραμείνουν τα στρατεύματα τη Αρμενίας εντό του Ναγκόνο Καραμπάχ, μόνο μα ενδιαφέρει από τι γύρω περιοχέ να φύγουν. Γιατί άλλαξε αυτό. Η ομάδα του Μίσκ είπε επιστροφή από τη επιστροφή των γύρω του Ναγκόνο Καραμπάχ περιοχών στην, στο Αζερβαϊτζάν. Αυτή είναι η διατύπωση της ομάδας του Μίνσκ και δεν λέμε εμείς τίποτα διαφορετικό. Οπότε για τον Αγκόνο Καραμπάχ υπάρχει το θέμα του νομικού καθεστώτος μέσω μιας νομικά δεσμευτική έκφραση της ελεύθερης βούλησης του λαού. Αυτό θα πρέπει να γίνει με την παροχή ε, διεθνών εγγύσεων και επιχειρήσεων διασφάλιση της ειρήνης. Αυτά λέει ε, κατά γράμμα το πρωτόκολλο του Μίνσκ. Δηλαδή αντιφάσκουμε σε σχέση με το ψήφισμα του 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ίσως ήταν λάθος. Ναι, όντως είναι το κείμενο αυτό του, της ομάδας του Μίνσκ και, και πιστή η αντιγραφή. Αλλά έχει δίκιο και συνάδελφος, γιατί αν ε, οι σκιώδεις ηγητές ε, κατέληξαν σε αυτή τη συμβαστική λύση και αν τελικά μπορέσουμε να διαγράψουμε από τις γύρω κατεχόμενες περιοχές, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι και να είμαστε και λίγο πιο φιλόδοξοι από την ομάδα του Μίνσκ. Πάντως, αν συμφωνήσουν ε, οι συνάδελφοι του ΕΛ και των άλλων ομάδων να, να διαγράψουμε τις τελευταίες λέξεις and surrounding occupied ε, regions, δεν έχω πρόβλημα. Θα προχωρήσουμε και λίγο περαιτέρω από τη διατύπωση του Μίνσκ. I am the shadow. I, I wanted I wanted to make this Ήθελα να κάνω αυτή την πρόταση να συζητήσουμε σήμερα τις δύο εκθέσεις με τους ε, σκιοδησίτες και να φύγει η λέξη surrounding από την συμβαστική υπαριθμό 6 της Αρμενίας και την 2 του Αζερβαϊτζάν. Θυμάμαι επίσης πως είχα κάποιες επιφυλάξεις αλλά μάλλον δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε στις συναντήσεις των σχεδόν. Δεν νομίζω. Καλά. Ε, εν πάση περιπτώσει είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι η ομάδα του Μίνσκ. Πρέπει να πούμε αυτά τα οποία έχουμε στο τελευταίο ψήφισμα. Να το ξεκαθαρίσω. Ο συμβιβασμό ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο-τριών ομάδων. Η ομάδα μου δεν συμμετείχε. Και ζητήσαμε μία άλλη συνάντηση για να καταλήξουμε. Αλλά συμφωνώ. Η Άννα έχει δίκιο. Αυτά υπάρχουν ήδη αλλού. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση. Σας ζητάμε να εξηγήσετε γιατί να μην ε, αποσυρθούν οι αρμενικές δυνάμεις από όλες τις περιοχές. Ε, μας είπατε γιατί είναι η διατύπωση του Μίνσκ. Μα ο λόγος ποιος είναι. Το επιχείρημα. Τα έγγραφα του ΟΗΕ περιέχουν την έκφραση όλες τις περιοχές. Πείτε μου το λόγο, γιατί τους ζητάμε να μείνουν εκεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι θα ήθελα να πω συναδέλφους η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή μας ε, δεν θα πρέπει να συμπεριφέρεται ως Σταύρος ε, ενιαλοπολείο και να προκαλέσει ε, περισσότερες ζημιές στην όλη διαδικασία. Η εντολή, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εντολή του ΟΑΣΕ είναι στους συμπροέδρους της ομάδας του Μίνσκ, που διαπραγματεύτηκαν τώρα, άμα μας αρέσει, δεν μας αρέσει, υπάρχουν, πλευρέ, υπάρχουν προβλήματα με τις αρχές του Μίνσκ, αλλά αυτολεξί περιέχονται στη διακήρυξη της Μαδρίτης αυτές οι αρχές. Αν θεωρούμε πως έχουμε κάποιο άλλο μέσο για να πιέσουμε και τις δύο πλευρές, να το κάνουμε, αλλά νομίζω πως θα κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά ε, παρά καλό στη σύγκρουση αυτή. Και επιμένω εγώ να μείνουμε στη διατύπωση που υπάρχει στη συμβαστική λύση 6, ιδίως στην άλλη έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Arvoisa puheenjohtaja, I say now. Θα... θα τα πω φιλανδικά. Όπως ε, θα διαπιστώσατε, το βασικό πρόβλημα είναι η συμβιβαστική υπαριθμών 2 της έκθεσης για την, το Αζερμπαϊτζάν που είναι η, το, η ίδια συμβιβαστική λύση με την ε, υπαριθμών 6 της έκθεσης για την Αρμενία. Και θα πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με τον πρόεδρο Μπροκ ότι θα μπορούσαμε τελείως να αφαιρέσουμε το Βόρειο Καραμπάχ από αυτό το κείμενο. Εχθές αποφασίσαμε στην τροπολογία τη Συμβαστική 2 για την έκθεση για το Αζερβαϊτζάν θα γινόταν μια ε, ψηφοφορία. Άρα λοιπόν για την αρχή είμαι υπέρ και στη συνέχεια από εκεί που λέει are linked to συνδέονται με πιστευτές, με αξιόπιστες δεσμεύσεις για ουσιαστική πρόοδο είμαι κατά. Η ομάδα μας δεν είναι υπέρ αυτού του δεύτερου τμήματος λοιπόν και σας καλώ να αφαιρέσετε την αναφορά στο Βόρειο Καραμπάχ στο δεύτερο εδάφιο της συμβαστικής στο δεύτερο τμήμα μάλλον της συμβιβαστικής τροπολογίας, γιατί βλέπετε ότι δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και δεν θέλουμε εδώ να θέξουμε αυτήν, την, ε, αυτό το θέμα. Αυτή είναι η δουλειά της ομάδας του Μίνσκ. Αυτή πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα και ακόμα και αν στο κοινοβουλίο θέλουμε να κάνουμε σωστά πράγματα, δεν νομίζω πως εμείς είμαστε σε θέση να λύσουμε το πρόβλημα. Η συμβαστική 2 λοιπόν της έκθεσης για το Ατζερβαϊτζάν. Το πρώτο τμήμα είναι ένα τμήμα το οποίο θα στηρίξουμε. Μπορώ και να το διαβάσω αν έχει την καλοσύνη ο κύριος Μπρόκ να με ακούσει. Προτείνω κατά τμήματα τροπολογία για τη συμβιβαστική ε, τροπολογία. Και έχω βάλει θετικό πρόσημο στην αρχή αυτής της συμβιβαστικής και αρνητικό στο τέλος της ίδιας συμβιβαστικής. Στο τέλος αυτής της συμβιβαστικής βρίσκονται όλες οι δυσκολίες ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή την περιοχή, όμως ε, ανάλογα με την ομάδα και ανάλογα με τους σκεώδεις ε, θα δούμε τι θα γίνει. Και όλα τα άλλα θέματα είναι ίσονο σημασία. Αλλά για παράδειγμα, επίσης ανησυχώ για τις στατιωτικές δαπάνες. είναι τεράστια στο Αζερβαϊτζάν. Αλλά υπάρχει και άλλη πτυχή. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες της Ένωσης πουλούν όπλα. Γιατί το κάνουν αυτό. Επίσης συμφωνώ με την κυρία Λούνα Τσέκ να, να στείλουμε έναν ειδικό απεσταλμένο για να ερευνήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα Δεν ξέρω ποιος θα αποφασίσει για το δημοψήφισμα, αλλά είχε γραφτεί αυτό στα προηγούμενα έγγραφα τα φετινά. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ εδώ τον εισηγητή της ομάδας μου για τη συμβεστική τροπολογία 6. Αντιστοιχεί σε δύο τροπολογίες έκθεση για την ΜΑΚΙ. Δεν συμφωνώ με την τροπολογία αυτή αλλά θα μπορούσαμε να διαγράψουμε κάθε αναφορά στα κριτήρια της ομάδας του Μίνσκ και να μιλήσουμε απλώς για τις γενικές αρχές ε, της ομάδας του Μίνσκ και της συνεδρίασης της Ακούιλα. Ε, σέβομαι τους κυρίους ε, Κούκαν και Μπρισάτζιτς, αλλά η αντίστοιχη διατύπωση του ΟΗΕ ήταν πριν από 20 χρόνια όταν δεν υπήρχε καμία προοπτική για, την, για τον διακανονισμό της κρίσης και τότε η, παγκόσμια, η ε, παγωμένη αυτή συγκρούση ήταν σε έκριθμη κατάσταση ενώ η ομάδα του Μίνσκ είναι πιο ρεαλιστική και προσπαθεί να ε, βρει μια λύση με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν. γνωρίζουμε ότι τα σύνορα και τα διεθνή σύνορα ε, στην πορεία της ιστορίας διαμορφώθηκαν με πολύ διαφορετικό τρόπο και θα πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό με βάση την πολιτική βούληση γιατί αν να ξεπεράσουμε κάποια όρια τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί. Ο κύριος Βάιγκλ ζήτηση για απόσυρση των ε, αραδαπών στρατευμάτων από την Αρμενία. Με αυτό θα υπονομεύσει την ασφάλεια της ίδια ε, ίδιας Αρμενίας. Είναι σαν να λέμε να αποσύρει τα στρατεύματά του, ε, να αποσύρει στρατεύματά του από τις βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Δεν συμφωνώ. Όπως είπαν ο Μπροκ, Τζολάιν και άλλοι, ε, για τις τροπολογίες της ε, κυρίας Λούνατζεκ είμαστε υπέρ της τροπολογίας 72, ε, αλλά όχι υπέρ της 108 και της 78. Πάντως το βασικό ζήτημα είναι οι συμβαστικές τροπολογίες 6 και 2. Είναι ένα πακέτο αυτές οι τροπολογίες, είναι ο μοναδικός τρόπος για να σημειώσουμε πρόοδο και δεν έχει κανένα νόημα να φιλοδοξούμε, να ξεπεράσουμε την εντολή της ομάδας ε, του Μίνσκ και τη διατύπωση αυτής της ομάδας. Ήταν πολύ έξυπνη η διπλωματική προσπάθεια της ομάδας του Μίνσκ τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι να το ξεπεράσουμε. Ήταν, θα ήταν ε, ανόητη μια τέτοια προσπάθεια και συμφωνώ με την κυρία Γετερμάκη να ε, εμείνουμε στη διατύπωση αυτή είτε να τη δεχτούμε ως πακέτο, ως σύνολο ή αλλιώς να μην αναφέρουμε τίποτα απολύτως. Ευχαριστώ. Τώρα έρχομαι στην τελευταία μου παρατήρηση. Θα προσπαθήσω να μιλήσω με τους δύο συγητές, ίσως και τους δύο συγητές, σήμερα το απόγευμα. Δεύτερον, αν δούμε το στρατικό προλογισμό μίας από τις δύο χώρες, είναι όσο ο προπολογισμό τη άλλη χώρα ολόκληρη. Με την ανάλογη αύξηση. Ε, κάνα δύο φορέ ήμασταν στα όρια του πολέμου. Και οι αρχές του Μίνσκ βοήθησαν να οριστεί ένα πλαίσιο έτσι ώστε κανείς να μην έχει άλοφη να ξεκινήσει πόλεμο. Σκεφτείτε το αυτό. Θέλω να αποφύγω η γνωμοδότηση να οδηγήσει τη μία ή την άλλη πλευρά να ξαναξεκινήσουν. Τα τελευταία δύο χρόνια ήμασταν στα όρια του πολέμου. Δεν είναι πράγματα αυτά για να παίζουμε Παρακαλώ λοιπόν να το συζητήσουν ξανά οι ομάδες και να το λάβουν υπόψη για, τις, ε, ε, για τους καταλόγους ε, ψηφοφορίας. Στρατιωτικά μιλώντας είναι μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές, το ανέφερε ο κύριος Λαντσμπεργκης, με επιρροή κάποιου ο οποίος αγοράζει όπλα και τα δίνει στον άνθρωπο. Ε, έτσι γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι στο συμφέρον της Ευρώπης. Μιλάμε για τον βόρειο γείτονα εκεί της περιοχής. Λάβετε το υπόψη, δεν πρέπει να δώσουμε άλοθη σε μία από τις δύο πλευρές να φύγει από το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί. Δεν είμαστε το μακρύ χέρι της μίας ή της άλλης κυβέρνησης εδώ πέρα. Νομίζω πως ξέρω για τι πράγμα μιλάω. Και έτσι, ε, συμβαστική λύση η οποία προτάθηκε είναι σωστή και δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κομμάτια από αυτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Σπάνια λέω πράγματα έτσι, τόσο σοβαρά. Σπάνια. Αλλά εδώ πέρα ξέρω τι λέω. Και λάβετε το υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε σημείο 7, λοιπόν. Ο κύριος Χάουιτ. Mr. Κύριε Χάουιτ. Um, Συγγνώμη Πρόεδρε, νόμιζα πως ε, αναφερόσασταν σε μένα ε, λόγω του θέματος της ημερήσιας διάταξης και ότι δεν μου είχατε δώσει ακόμα το λόγο. Είναι κάπως δύσκολο να μιλήσει κανείς. Μπορείτε να ζητήσετε ε, να γίνει λίγη, λίγο ησυχία. Πρόεδρε, παρακαλώ, μπορείτε να ζητήσετε να γίνει ησυχία στην αίθουσα. Τα καταφέρατε εσείς ο ίδιος. Το χιούμορ σας βοηθά σε αυτές τις περιστάσεις, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ένα θέμα το οποίο θα είναι λιγότερο επίμαχο σε αυτή την ε, επιτροπή από το προηγούμενο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει προετοιμαστεί από την ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ε, θα ήθελα εξ αρχής να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν εκεί για τη συνεργασία τους. Το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας ε, στην Επιτροπή, αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας, αυτό που θέλω να κάνω είναι να εστιάσω την προσοχή στα βασικά θέματα της έκθεσης, τους τομείς ε, όπου μπορούμε να κοινοτομήσουμε και τις νέες ιδέες, αν και φυσικά ευχαρίστω θα απαντήσω σε οποιαδήποτε περαιτέρω ερωτήματα ή παρατηρήσεις για τις συμβιβαστικές ή για τις συγκεκριμένες τροπολογίες των συναδέλφων συναδέλφων κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Επίσης θέλω να πω εισάγοντα αυτή την ε, παρουσίαση ότι όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα χρονοδιαγράμματος και τη διαδικασία, όχι προβλήματα του ίδιου του Κοινοβουλίου, αλλά προβλήματα στο πλαίσιο τη υπηρεσίας Εξωτερική δράση και του Συμβουλίου. Και εξ αρχής θα πω ότι είμαι ευτυχής πως όλα αυτά τα έχουμε εμείς ξεπεράσει και μπορέσαμε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και να πω ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ήταν πολύ σαφής, έμαθαν από τις δυσκολίες του περασμένου χρόνου και τις αντιμετώπισαν. Επίσης έγιναν ε, σε πολύ ε, σημαντικές εκθέσεις σε αυτή την Επιτροπή ε, την έκθεση για το εθνικό για, για το μάλλον Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Ντόφλερ, ε, Κράισερ επίσης η έκθεση για τα υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κυρίας Χάουτελα και φυσικά οι εργασίες για το κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα Όλα αυτά είναι αναφορές για την εκθεσή μου. Τα βασικά του συμπεράσματα τα έχω υιοθετήσει. Θέλω μόνο να εφαρμοστούν και όχι να συζητήσουμε περαιτέρω αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους ε, για τη δουλειά που έκαναν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα στο οποίο κινούμεθα. Ε, στην παράγραφο 84 αλλά και αλλού γίνεται λόγος για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μάθει τα μαθήματα από τις στενές της σχέσεις με τα αυταρχικά καθεστώτα, λαμβάνοντας, αναφέροντας το παράδειγμα της ε, Λιβύης και δεν σημαίνει μόνο ότι θα πρέπει να μάθουμε από τα παλιά μας λάθη, αλλά θα πρέπει να εμποδίσουμε την επανάληψη παρόμοιων λαθών στο μέλλον. Ε, επίσης θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι προκλήσεις των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων να θέλουμε πραγματικά να επηρεάσουμε και τα όσα γίνονται εκτός και τονίζω ιδιαίτερα τα θέματα του ασύλου και των εκτάκτων μεταγωγών και θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα. Έχουμε επίσης στην παράγραφο 4 όπου ζητάμε επιτάχυνση της διαδικασία ε, για την ε, πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαμαρτυρόμεθα για τις ε, καθυστερήσεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ε, Επίση, θα ήθελα να πω σε όλου του συναδέλφου τη Επιτροπή ότι θα είναι ο πρώτο ειδικό ε, εκπρόσωπο για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ο Χαβιέ Σολάνα ήταν ένας προσωπικός εκπρόσωπος, είναι ένα επίτευγμα το ότι το ζητήσαμε από την είπατε εκπρόσωπο και έχουμε επιμείνει για τα προσόντα, την εμπειρία και τα καθήκοντα που θα πρέπει να αναλάβει ο δικός μας εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην παράγραφο 35 για τις εμπορικές συμφωνίες μιλάμε για τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διαπραγματεύσεις και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχετική ρήτρα, ανθρώπινα δικαιώματα και η κατάσταση προόδου τους μετά από την εφαρμογή, καθώς και η ρήτρα που θεσπίζει ένα μηχανισμό για αναστολή αλλά και περιγράφει τα βήματα στα οποία, ε, τα οποία οδηγούν στην αναστολή, παράγραφοι 14 και 15. Παράγραφος 16 κάνει λόγο για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δουλειάς της στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνεργασία με τρίτες χώρες, υποβολή συστάσεων, αναχώρα ε, στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στη στρατηγικά μας έγγραφα για τις τρίτες χώρες. Στην παράγραφο 28 γίνεται λόγος για ένα θέμα το οποίο συχνά έχουμε αναφέρει, την παρακολούθηση δηλαδή ε, και τη συνέχεια που δίνεται στις ε, ειδικές τακτικές αποστολές παρατήρησης δύο χρόνια μετά από την ε, ολοκλήρωση της αποστολής. Επίσης αναφέρουμε επικρίσεις όσον αφορά την έλλειψη προόδου στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην παράγραφο 31 και λέμε ότι πολλές φορές ε, αποφεύγεται ο έλεγχος και η παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους ε, πριν προβεί σε τέτοιου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι θα πρέπει η κάθε ομάδα εργασία να καταλήγει σε συμπεράσματα. Επίση, επιστήνουμε την προσοχή στο γεγονό ότι η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, κατά τη γνώμη μα, Ε, δεν ε, αξιοποιεί καταλήλως και με διαφανή τρόπο τον ε, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε τώρα επίσης ένα αίτημα για μια μεγάλη πρωτοβουλία για τις χώρες κατά των βασανιστήριων. Δεν έχουν συνυπογράψει αρκετές χώρες και θα πρέπει αυτό να είναι βασική μας προτεραιότητα στην πολιτική γυπνίασης. Στην παράγραφο 55 τώρα Αναφέρουμε την συμφωνία στον δημοσιονομικό κανονισμό μετά από το 2014 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα έγγραφα για στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι συγκεκριμένα δεν θα είναι ε, έγγραφα κατεξουσιοδότηση, για κατεξουσιοδότηση πράξης και όλοι γνωρίζουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον τρόπο με τον οποίο στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, δαπανά τα χρήματά της. Περίγραφη, παράγραφη 59 με 62 θυμίζουμε το γεγονός ότι φέτος ήταν η επέτειος ε, του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια των γυναικών ε, και θέλουμε, μάλλον ζητούμε ο κανονισμός σχετικός να υιοθετηθεί σε όλες τις αποστολές και να, να υλοποιηθεί ε, για την καταπολέμηση της βίας κατά των ε, γυναικών μέσα σε όλα τα στρατιωτικά σώματα και όλες τις ειρηνευτικές δυνάμεις. Επίσης, ε, επαναλαμβάνουμε την, ότι είμαστε κατά των αναγκαστικών γάμων. Παράγραφη 68 με 72 για πρώτη φορά νομίζω σε μια τέτοια ετήσια έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου μιλάμε για το ίντερνετ, ε, τα κοινωνικά μέσα και ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταδικάζουμε την ε, λογοκρισία των καταπιεστικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων. Επίσης για το θέμα των ε, επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, της επιχειρηματικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνουμε, στηρίζουμε το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει συμφωνηθεί ε, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μάλιστα έχουμε δύο φορές δει τον καθηγητή του οποίου έργο είναι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι δικαιωμάτων Επίσης έχουμε μιλήσει, μιλάμε για την εφαρμογή της μελέτης του Εδιμβούργου για το πώς μπορεί κανείς να κλείσει τα κενά διακυβέρνησης μέσα στην Ευρώπη για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, πράγμα το οποίο σε, καλύπτεται σε μάκρος από την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τέλος, στις τελευταίες παραγράφους μέχρι την 98 μιλάμε για τη στρατηγική αναθεώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ξέρετε ότι υπήρξε μια συμβαστική στην υποεπιτροπή που είπε ότι θα χρησιμοποιήσουμε την ετήσια έκθεση ώστε να συμβάλλουμε χωρίς ε, αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα καταθέσουμε περαιτέρω ψηφίσματα από το Κοινοβούλιο και όλοι ακούσαμε χθε από τη Βαρόνη Άστον πως ε, είναι προσιλωμένη στην κοινοβουλευτική συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το τμήμα λοιπόν του σχεδίου ψηφίσματος υποστηρίζουμε όχι μόνο τον ειδικό εκπρόσωπο αλλά και την ομάδα εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα να, βασί... να εδρεύει στις και να συντονίζεται όπως κάνουμε για κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, και όχι να πηγαίνουν έρχονται από τις διάφορες πρωτεύουσε των κρατών μελών. Συγκεκριμένα συμπεράσματα επίσης θέλουμε μετά από κάθε ε, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία εστίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να υπάρχει κοινή βάση επίσης για τα έγγραφα που αφορούν τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να είμαστε συνεπείς και μιλάμε και για μια νέα σχέση με τις ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην τους βλέπουμε ως φορείς απλώς που ε, εφαρμόζουν την πολιτική αλλά ως εταίρους. Ζητούμε επίσης την ε, δημιουργία μηχανισμών όταν υπάρχουν ε, καταγγελίες για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μηχανισμοί που θα μπορούν να μας επιτρέψουν να τα αντιμετωπίσουμε σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και να παροτρύνουμε για την μεγαλύτερη κινητικότητα. Και επίσης ζητάμε συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ορισμένοι μπορεί να πούνε ότι θέλουμε περισσότερη επιρροή ω Κοινοβούλιο. Εγώ θεωρώ πως τμήμα αυτής της έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη, να δίνεται μάλλον μεγαλύτερη έμφαση στην λογοδοσία ε, της Ένωσης για το πώς προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω. Και αυτό είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και νομίζω πως ε, Ε, έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς καλύτερα τη δουλειά μας και να δημοσιοποιήσουμε περισσότερο αυτήν την λογοδοσία. Εγώ είμαι πολύ αφοσιωμένη σε αυτή την εργασία και ξέρω και πολλοί κόσμοι στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, με μεγάλο πάθος ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Παρακαλώ λοιπόν να υπάρξει συνένεση από όλες τις ομάδες όταν θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ο Θα ήθελα να επισημάνω ότι Έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία με αυτή την ετήσια έκθεση ένα πολύ διακεκριμένο έργο. Βέβαια, μιλάμε για την έκθεση του 2009 και ολοκληρώνουμε το έργο αυτό το 2012 καταρχήν. Κανονικά θα πρέπει να ολοκληρώνουμε τον ίδιο χρόνο τις εργασίες αυτές και σήμερα να ασχολούμαστε με την έκθεση του 2011 και όχι του 2009 αλλά διάφορες περιστάσεις έλαβαν χώρα και είχαμε και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, και της ΕΠΑ, της εκπροσώπου καθώς και του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά και την ε, ανάγκη για πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Από αυτή την άποψη η αιτήσια αυτή έκθεση είναι μια συνολική έκθεση και περιλαμβάνει κάποιες ε, γενικές παρατηρήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η τελική εκδοχή της αιτήσιας έκθεσης του κυρίου Χόουιτ είναι ένα πολύ αξιόλογο έγγραφο. Ε, κατατέθηκαν ε, γύρω στις 300 τροπολογίες, συντάχθηκαν και συμβιβαστικές τροπολογίες και χάρη στην αγαστή συνεργασία που είχαμε με τους συναδέλφους, καταφέραμε τελικά να συμπληρώσουμε την έκθεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις ε, ζητήθηκαν ψηφοφορίες κατά τμήματα και μπορούμε να συμφωνήσουμε και εκ μέρους του ΕΛΚ με τις συμβαστικές τροπολογίες όλων το, με όλες τις τροπολογίες, με εξαίρεση βέβαια κάποια εδάφια που θα καταψηφίσουμε στα πλαίσια των ψηφοφοριών κατά τμήματα που ζητήσαμε. Ε, γίνεται ένα είδος συστηματοποίησης στην έκθεση αυτή, ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιπτώσεις ανθρω... ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως μας εξήγησε και ο εισηγητής. Ε, επίσης, με την ετήσια αυτή έκθεση καταφέραμε για την πλειονότητα των περιπτώσεων να καταλήξουμε σε συμφωνία προκειμένου να ε, δημιουργηθεί μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης, χάρη και συμβαστικές ε, προτάσεις. Τελικά, εκεί που δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα υποβάλω τρεις προφορικές τροπολογίες. Η πρώτη είναι πολύ σύντομη αφορά κάποια θέματα σύνδεσης, εκεί που μιλάμε για, κάποιες, ε, για κάποια σημεία της έκθεσης της κυρίας Άστον και το θέμα της κοινωνίας των πολιτών μαζί με το Ταμείο ε, της ε, Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε αυτή η πρόταση ως κοινή και καλό θα ήταν να αναφέρουμε ρητά στις συμβαστικές τροπολογίες ότι τα θέματα της δίωξης των χριστιανών στον κόσμο είναι κάτι που θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά στην έκθεση, να λαμβάνεται υπόψη και στις συμβαστικές τροπολογίες, να αναφέρεται ρητά. Γιατί μιλούμε για τη δίωξη θρησκευτικών μειονοτήτων. Αλλά με την, με την έκριση του ψηφίσματος για την Ιγυρία, δεχτήκαμε την ειδική μνήμη της δίωξης των χριστιανών. Κάτι αντίστοιχο θέλουμε με την προφορική αυτή τροπολογία να προσθέσουμε και στις συμβαστικές ε, προτάσεις της έκθεσης ε, του κ. Χόουιτ. Η Αραβική Άνοιξη μας έδειξε ότι μερικές φορές ε, οι εξελίξεις μετά την Αραβική Άνοιξη, είδαμε τι έγινε με την κοπτική κοινότητα στη, στην Αίγυπτο, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Δηλαδή, περιμένω μια καλύτερη τήρηση των προδιαγραφών και σεβασμό των θρησκευτικών κοινοτήτων, κάτι που δεν έγινε πάντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τελευταία θανατική ποινή στη Λευκορωσία. Όλοι συμφωνούμε ότι των ποινών η θανατική ποινή δεν θα πρέπει να εκτελείται και ακόμη και να προβλέπεται στην ένωμη τάξη δεν θα πρέπει να εκτελείται. Κανονικά θα έπρεπε να μην εφαρμόζεται πουθενά, να απαγορεύεται, αλλά υπάρχουν ακόμη ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή. Ακόμη και οι ελάχιστες προδιαγραφές για τα οικογενειακά δικαιώματα, ε, για την ταφή των καταδικασμένων, ούτε καν αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη από ορισμένε χώρες και αυτό είναι πραγματικά ελάχιστη προϋπόθεση, ελάχιστη προδιαγραφή. Γι' αυτό και θα υποβάλω μια προφορική τροπολογία με αυτό το περιεχόμενο, ώστε αυτές οι ελάχιστες προδιαγραφές να τηρούνται ακόμη και σε περίπτωση ε, εκτέλεσης θανατικής ποινής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έξι λεπτά είχαμε πει. Λοιπόν, ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά καλά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε για την έκθεση αυτή. Εγώ ήμουν σκιώδης ηγητής και αισθάνθηκα ιδιαίτερη χαρά και τιμή α, για τη συμμετοχή μου σε αυτή την έκθεση. Είμαι και μέλος Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια. Η έκθεση είναι περιεκτική, α, ισορροπημένη, αξιόλογη και λαμβάνει υπόψη και πολιτικές και ηθικές ευαισθησίες. Κάτι είναι πολύ σημαντικό και όταν ερμηνεύουμε μερικά ευαίσθητα θέματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα και καταστρατηγήσεις τους, είναι δύσκολο μερικές φορές να βρούμε ελάχιστο κοινό παρανομαστή, γιατί διαφέρουν οι προσεγγίσεις μας. Πάντως η, ισχύ και η αξία της έκθεσης αυτής, εκτός από τη διαδικασία συνεργασίας, ήταν και το γεγονός ότι μας επέτρεψε να συζητήσουμε πολλά θέματα και να λάβουμε υπόψη όσο το δυνατό περισσότερες απόψεις. Η σε αυτή η έκθεση θέλει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πια ένα είναι ο επίσημος πολιτικός λόγος της Ένωσης και μάλιστα κοινό λόγος ε, από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Και νομίζω ότι ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο συνδετικός ιστός της ε, δημοκρατίας. Θα πρέπει λοιπόν να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου και κατά των απολυταρχικών καθεστώτων, αυταρχικών καθεστώτων σε περίπτωση που διαπιστώνουμε καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια, κανένα κράτος, όσο δημοκρατικό και αν είναι και όσο ελεύθερο, δεν μπορεί να θεωρεί ότι υπερέχει της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή της ανθρώπινης ζωής. Γιατί η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια δεν είναι η ανθρωπινη ζωη και αξιοπρεπεια δεν ειναι ιδιοκτησια του κράτους. Και με τέτοιες σημαντικές εκθέσεις ε, υπενθυμίζουμε την πολύ αυτή σημαντική αρχή, κύριε Πρόεδρε, που από ό,τι ξέρω είναι κοινή αρχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και την εστερνίζονται όλα τα κόμματα. Επαναλαμβάνω, αισθάνθηκα μεγάλη χαρά για την ευκαιρία συνεργασίας που είχαμε με τον κύριο Χόουιτ και νομίζω ότι καταφέραμε όσα μπορούσαμε με την έκθεση αυτή. Βέβαια κάποιες εκκρεμότητες έχουν παραμείνει γιατί καμία έκθεση δεν πρόκειται ποτέ να καλύψει αυτό το τεράστιο φάσμα, αυτό το τεράστιο πεδίο που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά έχοντας υπόψη τις συζητήσεις ε, και την έκθεση, πιστεύω ότι είναι δίκιο να πούμε ότι είναι πολύ επίκαιρη αυτή η έκθεση και πολύ αξιόλογη. Ευχαριστώ. Thank you, like... Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, τον συζητητή και τους σκιώδες για την φανταστική δουλειά τους. Είναι ωραίο αυτή η έκθεση. Ισορροπημένη και με ουσία όμως, με προτάσεις ε, ε, που πραγματικά καθιστούν σαφές πως ε, θέμε αυτό το νήμα που ενώνει την πολιτική μας που λέει η κυρία Άστον αλλά να είναι πραγματικά μέρος της πολιτικής ένωσης από την ενέργεια, στο εμπόριο, την ανάπτυξη όπου χρειαζόμαστε μία ενιαία προσέγγιση και τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι ε, Επειδή λοιπόν και εγώ έχω καταθέσει κάποιες ε, τροπολογίες για κάποια πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν, είμαι ικανοποιημένη με τη δουλειά του Ρίτσαρντ Χάουιτ, ε, του εισηγητού και των σκιωδών εισηγητών. Πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Ε, επίσης για το Ταμείο το Ευρωπαϊκό για τη Δημοκρατία πράγματι πρέπει να είναι υπό την εποπτεία του Κοινοβουλίου και να μην είναι γραφειοκρατικό και δεν θα πρέπει να αφαιρεί κονδύλια υφιστάμενα αλλά να προσθεθούν και άλλα. Επίσης για τις εκλογές, γιατί λεφτά από τα μέρος των χρημάτων από αυτά τα οποία εξοδεύουμε πάνε σε εκλογές, αλλά πρέπει να φροντίσουμε πως οι εκλογικές διαδικασίες που παρατηρούμε ε, τελικά προωθούν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και όχι να νομιμοποιήσουν αυταρχικούς ηγέτες. Και βεβαίως ε, οι πολύ σημαντικές συνεισφορές που υπάρχουν για τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, να είναι μέλος, μέρος των μελλοντικών εκθέσεων, το τι γίνεται για τους αυτόχθονες αλλά και τις μειονότητες και βεβαίως η στρατηγική αναθεώρηση ε, του μηχανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ναι. Πολύ θετικές προτάσεις ε, και νομίζω πραγματικά πως ε, έτσι θα αποτελέσει τη βάση για τη δουλειά μας στο, στο μέλλον. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι βεβαίως ποτέ δεν έχουν εξαντληθεί αυτά τα ζητήματα αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα υπόδειγμα ε, και για το μέλλον και ε, όχι μόνο για την ανάλυση του παρελθόντος. Ευχαριστώ. Uh, um, ε, σύντομα, κύριε Πρόεδρε, η ομάδα μας γενικά στηρίζει την έκθεση Χάουιτ. Έχω συνεργαστεί με τον Ρίτσαρντ Εψηρά ετών για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα στηρίξουμε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες, όπως το μέρος δεύτερο της τροπολογίας 1, που καταδικάζει υπερβολικά κάποια κράτη-μέλη κατά την άποψή μας. Επίσης αποχή στην ε, τροπολογία 11 γιατί είναι πολύ ε, άκαμπτη σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Στην 23 θα υποβάλουμε προφορικές τροπολογίες ε, για να υποστηρίξουμε την θέση του σκιώδου συζητού του ΕΛΚ για τις αρχαίες χριστιανικές κοινότητες όπως οι κόπτες στη Μέση Ανατολή που αντιμετωπίζουν απειλή για την ύπαρξή τους εάν οι σαλαφιστές καταλάβουν την εξουσία στη συμβαστική υπαριθμό 18 για τη θανατική ποινή και την υπαριθμό 31 για τις ε, εκτρώσεις η ομάδα μου παραδοσιακά έχει ψήφο κατά συνείδηση Αυτή είναι η θέση λοιπόν των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Χάουιτ για την έκθεσή του. Εγώ είμαι συντάκτης γνωμοδότησης της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Χάουιτ και τα υπόλοιπα μέλη της ΑΦΕΤ να λάβουν υπόψη τις συστάσεις της γνωμοδότησης της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης. Στόχος είναι οι στάσεις αυτές να ακολουθούν και να ευθυγραμμίζονται με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας και να έχουμε μια συνεκτική εξωτερική πολιτική. Η ανακοίνωση για τις αρχές της δημοκρατίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει να διαπερνά όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η ολοκληρωμένη στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα όντω να διέπει όλες τις πολιτικές και να λαμβάνεται υπόψη. Θα ήθελα να ζητήσω μία ε, δημοσιονομική υποστήριξη που θα εξαρτάται και από την ε, τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο λεπτομεριακά κριτήρια για την ε, χορήγηση κονδυλίων σε τρίτες χώρες που να εξαρτώνται από την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές διανύουμε ούτως ή άλλως μια οικονομική κρίση, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί στήριξης της δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων, γιατί είναι το πιο από το μέσο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εξασφαλίσει καλύτερη συμπερίληψη του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διάλογο με τις τρίτες χώρες και ιδιαίτερα στα θέματα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Όλμαρ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Ρίτσελ Χάουιτ και αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω δύο από τα ευρύτερα ζητήματα που τον απασχολούν εδώ πέρα. Μου φαίνεται πως η συνέπεια θα έχει μεγάλη σημασία για την πολιτική αυτή, όπως επισημαίνει Ρίτσαρντ. Στα ανθρώπινα δικαιώματα Διάβασα πρόσφατα μία εκθεσή για τις κυρώσεις και το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Συμβούλιο για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρώ πως θα έχουμε αξιοπιστία μόνο αν υπάρχει εφαρμογή ομοιόμορφη. Το εάν θέλουμε τώρα να είμαστε φιλικοί με μια ξένη κυβέρνηση ή όχι είναι διαφορά. Αν κοιτάμε παραδείγματο χάρη τη Μέση Ανατολή, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρε όπω η Συρία ή και η Αίγυπτος και να μην λέμε τίποτα για τη Σαουδική Αραβία. Θεωρώ πως εδώ πέρα μπορούμε να δεχτούμε από τους Αμερικανούς ε, αν δούμε παραδείγματος χάρη ε, το νομοσχέδιο του Σεργέη Μαγκνέτσκι περί κράτους δικαίου και το πώς προσπαθούν ε, ένα συγκεκριμένο περιστατικό να το αντιμετωπίσουν νομίζω πως αυτό το παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για εμάς για την πολιτική μας και υπ' αυτή την έννοια όπως είπατε η ένταξή μας στην ΕΣΔΑ είναι κάτι το σημαντικό και λυπούμε για το ότι δεν επιθυμούν διάφορα καθεστώτα του, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία να το κάνουν αυτό. Πρέπει να μας στηρίξουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, πρέπει να συζητάμε τα... όχι μόνο αυτά τα οποία συζητήσαμε χθε με την κυρία Άστον, το τι κάνουμε εξωτερικά, αλλά και ο πιθανός ρόλος ε, του ειδικού απεσταλμένου για να εργαστεί εσωτερικά στις υπηρεσίες κομισιών, να εκπαιδεύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να ενσωματώνει την πολιτική αυτή και γενικώ ε, να αυξάνει την ικανότητα της Ένωσης ε, να ασχοληθεί αποτελεσματικά με αυτά τα ζητήματα. Ελπίζω επίσης πως ε, η ύπατη εκπρόσωπος θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να βρει ζητήσει μεγαλύτερη στήριξη ε, για να ασκήσουμε πίεση στις ΙΠΑ για να ενταχθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παραδείγματος χάρη να κυρώσουν τα πρωτόκολλα καθώς αυτή τη στιγμή το δικαστήριο δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο θα μπορούσε και προφανώς δεν έχει αρκετή στήριξη. Εξαγωγέ όπλων όπως επισημαίνει ο εισηγητή, είναι πολύ σημαντικές και συμφωνώ απολύτως. Πως ε, η περαιτέρω προσοχή στην εφαρμογή της κοινή θέση του 2008 στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς ε, πολλές παραβιάσεις δεν θα μπορούσαν να διαπραχθούν χωρίς τα όπλα που πουλάνε κρατημέλη ανά τον κόσμο και έχω την εντύπωση πως η στήριξη των τριών θεμάτων της είπα της εκπροσώπου για συλλογική δράση θα επιτρέψει στην Ένωση στο πλαίσιο της συνολικής της πολιτικής να έχει συγκεκριμένα σημεία έμφασης ε, σε ζητήματα που μας ανησυχούν και στο μέλλον ε, θα μπορούμε να είμαστε πολύ πιο ε, ενημερωμένοι και ευθυγραμμισμένοι με τις εξελίξεις της παγκόσμιας. Συνελώνται λοιπόν να συγχαίρουμε τον εισηγητή και συμφωνούμε με την έκθεση αυτή. Να πω κάτι γρήγορα για εξ της ομάδας μας, το οποίο μου θύμισε ο Γκράχαμ. Παράγραφος παριθμών 4, η οποία, και αυτό είναι κάπως ασύνηθες και ηρωνικό, καθώς είναι ο συντάκτης Βρετανός, ασκεί κριτική στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την ε, ένταξη της Ένωσης ε, στην ΕΣΔΑ. Ε, έχουμε υποβάλει τροπολογία να διαγραφεί αυτό το κομμάτι. Ξέρω πως το κόμμα του Γκρέμ και το δικό μου κόμμα είναι στην κυβέρνηση συγκυβερνούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εδώ πέρα διαφωνούμε, καθώς επί της αρχής είμαστε κατά η συντηρητική. Ξέρω πως τώρα βεβαίως είναι υποχρέωση από τη συνθήκη, αλλά είναι μια συνθήκη την οποία, στην οποία ήταν κατά το δικό μου το κόμμα. Και θεωρούν πως έτσι θα δημιουργηθεί σύγχυση, αλληλεπικάλυψη, προβλήματα αρμοδιότητας του ΔΕΚ και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Ντέβιτ Κάμερον μάλιστα πρόσφατα δεδομένου του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει να μεταρρυθμίσει το δικαστήριο καθώς εμείς θεωρούμε ότι το δικαστήριο μπαίνει στα χωράφια που δεν το σπέρνουν και ασχολείται με αποφάσεις ε, ερετών κοινοβουλίων όπως το δικαίωμα των φυλακισμένων να ψηφίζουν. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να περιγράφουμε Ρίτσαρτ τη χώρα μας ως χώρα η οποία φέρνει προσκόμματα. Ευχαριστώ. Καταπληκτική αυτή η Επιτροπή, γιατί μπορεί να διαφωνούμε, αλλά τουλάχιστον υπάρχει κατανόηση. Δεν νομίζω. Αν νομίζω ότι καλό θα ήταν να ακούσουμε κάποιον από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, γιατί αν έχει, υπάρχει εκπρόσωπος εδώ, καλό θα ήταν να τον ακούσουμε πριν λάβω εγώ το λόγο για να ολοκληρώσω. Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Καλώς, τότε να απαντήσω. Κύριε Ξύπ. Ε, όντω μίλησε για την καθυστέρηση και το χρονοδιάγραμμα. Συμφωνώ, είναι πραγματικά ατυχέ που είχαμε τέτοια καθυστέρηση και συζητούμε τώρα το 2012 ε, τη έκθεση του 2009. Αλλά δεν ήταν δικό μα το σφάλμα. Είχαμε διαδικαστικέ δυσκολίες που νομίζω ότι διορθώθηκαν τελικά. Πάντως ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ξύμπ ε, για τη συνεργασία που είχαμε και για το συνεργάσιμο πνεύμα που επέδειξε στις διαπραγματεύσεις. Πάντως ε, θα είδατε κι εσείς ότι ακριβώς ε, επειδή δεχόμενος πολλές τροπολογίες ομάδας ε, ήθελα να σας ευχαριστήσω και εμπράκτος για την υποστήριξη της ομάδας και για τη στενή συνεργασία που είχαμε. Συμφωνώ επίσης με αυτά που είπατε για, την εκτε... για τις εκτελέσεις στη Λευκορωσία. Σας ζήτησα να καταλήξετε σε μια διατύπωση, υποβάλλατε τροπολογία, συμφωνώ πλήρως και νομίζω ήταν πολύ σημαντική η συμβολή σας και σας ευχαριστώ θερμά. Σε ό,τι αφορά την... το Ταμείο για τη Δημοκρατία είναι κάπως παραληπτικό αυτό το σχόλιο, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό για την ομάδα σας. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να προτείνουμε μία διατύπωση που να λαμβάνει υπόψη την Δεν έχει ακόμη συσταθεί αυτό το Ταμείο. Ε, παρακαλώ συνεννοηθείτε με τη γραμματεία για να βρούμε τη σωστή διατύπωση. Η μόνη δυσκολία και η διαφωνία που έχω μαζί σας και θα το κατανοήσετε, γιατί και εγώ κατανοώ τις δικές σας δυσκολίες και ευαισθησίες, αφορά την συγκεκριμένη διατύπωση που ζητάτε για την δίωξη των χριστιανών στην συμβαστική τροπολογία 24. Οι συμβαστικές τροπολογίες 23 και 24 είναι νέες παράγραφοι στο κείμενο μετά από μεγάλο αριθμό τροπολογιών που έλαβα για την ανεξιθρησκεία και την ελευθερία θρησκευτική πίστης και λατρεία. Προσπάθησα να καλύψω στο δυνατό περισσότερες τροπολογίε. Πάντως διαπιστώνω ότι σημαντικό στόχο τη δική σα ομάδα, και άκουσα και τον κύριο Τάνοκ, είναι να ε, γίνει η ρητή μνήμα των διώξεων των χριστιανών. Και εγώ χριστιανό είμαι. Επί τη αρχή δεν διαφωνώ και σαφώς είμαι ε, κατά των διώξεων ε, εις βάρος των χριστιανών. Αλλά σε κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πάντα αυτό κάνω εκ μέρους της ομάδας και πιστεύω ότι και είναι τέτοιο προς, το όφελος, προς όφελος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μιλούμε για διώξεις, να αναφέρουμε τις διώξεις κατά των θρησκευτικών κοινοτήτων και να μην ξεχωρίζουμε μία από αυτές τη χριστιανική κοινότητα προκειμένου. Όντως, στο κατεπήγον για την Ιγυρία πέρυσι τον Απρίλιο είχαμε ειδική μνήμα και το θυμάμαι και το αναγνωρίζω τη συμβολή σας, αλλά τον Ιανουάριο με το ψήφισμά μας για την ανεξιθρησκεία καταφέραμε τελικά να καταλήξουμε σε μια διατύπωση που μιλούσε για τη δίωξη των χριστιανών, αλλά ε, ανέφερε και ένα κατάλογο όλων των θρησκευτικών διώξεων. Εξήγησε εκτενώς ε, τους λόγους για τους οποίους κατέληξα σε αυτή τη διατύπωση που πρότεινα και με κάθε σεβασμό απέναντί σας ε, σας προειδοποιώ ότι δεν θα συμφωνήσω με την προφορική σας τροπολογία. Ε, κύριε Ντόνσκης, ε, και εκείνο διαφώνησε, δεν υπάρχει συνένεση για το θέμα αυτό. Πάντως, πολύ ευχαρίστω να ξανασυναντηθούμε και σας παραπέμπω στο ψήφισμα του Ιανουαρίου του περσινού χρόνου. Πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια αποδεκτή διατύπωση για να συμφωνήσουμε όσο είναι εδώ περισσότεροι στο ψήφι, στην έκθεση αυτή. Αν ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Δεν έχω συγκεκριμένες απαντήσεις να σου δώσω. Σε ευχαριστώ για τη συμβολή σου ε, και ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Ντόσκης που πραγματικά ήταν εξαιρετικός ε, σκιώδης ηγετής και πολύτιμος ε, συνεργάτες, στους φίλους ε, και συναδέλφους, στο, στο φίλο και συνάδελφο κύριο Τάνοκ, που ζήτησε διαγραφή της ε, συνέχισης της εξεταστικής, της ε, εξεταστικής επιτροπής, της προσωρής επιτροπής μάλλον για τις παράνομες μεταγωγές. Τότε εγώ ήμουν κυβέρνηση και το κόμμα ήταν αντιπολίτευση όταν έγινε η, η επίκριση αυτή. Και τώρα με κατηγορεί για αντιβρετανό επειδή επισημαίνω ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι μία από τις δύο μεγάλες χώρες που είναι γνωστές σε όλους που εμποδίζει την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην ΕΣΔΑ. Πάντως έχουμε αγαστές σχέσεις εργασίας με τον κύριο Ντάνο, ακόμη και όταν διαφωνούμε, εμπροκειμένου όμως διαφωνούμε. Εγώ ανέκαθεν ήμουν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι υπέρ των συμφερόντων συγκεκριμένε χώρε. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που διαπιστώνονται, υπάρχουν υπόνοιε για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να, διαλευκαίνονται, να οι περιπτώσει. Γι' αυτό και δεν δίστασα να κατανομάσω και την Βρετανία εδώ. Σε ό,τι αφορά τη ε, κατασυνείδηση ψήφου, ελπίζω να συμφωνήσετε πάντως με τις τροπολογίες της συμβαστικές 18 και 21. Η τροπολογία 21, μάλιστα, κατανοώ βέβαια αυτά που είπατε, αλλά η τροπολογία 21 μιλούν για την ε, υγεία των γυναικών. Βέβαια, περιλαμβάνεται η αναπαραγωγική υγεία, αλλά η παράγραφος 21 δεν αφορά μόνο την άμβλωση, όπως είπατε, είναι γενικώ για την υγεία των γυναικών. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Ελπίζω να συμφωνήσουν και τα μέλη της ομάδας με την παράγραφο, παρά την ψηφοφορία κατά το δοκούν. Κύριε Πρέντα, η δική σας έκθεση ήταν η πιο διεξοδική γνωμοδότηση Επιτροπής. Θα μελετήσω ε, περιστατωμένο τις ε, προτάσεις σας. Τον ευχαριστώ πάντως θερμά και τον κύριο Πρέντα για την σημαντική του συνεισφορά. Τώρα, το ψήφισμα για τις κυρώσεις, κύριε Βότσον, που υποβάλλεται μετά την ε, έναρξη των εργασιών για την έκθεση, θα μπορούσαμε ίσως μέσω μιας προφορικής τροπολογίας να το λάβουμε υπόψη. Και εδώ απευθύνομαι στη γραμματεία να το ελέγξει. Ελπίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε κύριε Βότσον και με άλλους για να περιλάβουμε και ένα σημείο για τις κυρώσεις. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια σταδιακή προσέγγιση, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι όλα ή τίποτα. Θα ήθελα πάντως να ληφθεί υπόψη και το σημείο αυτό. Και τέλος, για τον εσωτερικό λόγο της ύπαντης εκπροσώπου, υπάρχει και εδώ ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Τώρα, ε, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο συμφωνώ ε, μαζί σας κύριε Βότσον. Υπάρχουν πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν συμφωνήσει πλαίσιο ε, για συμφωνία και εφαρμογή των, ε, των αποφάσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και μάλιστα δεν, έχουν κυρωθεί, δεν έχει κυρωθεί η σύμβαση αυτή. Μάλιστα περιλαμβάνεται μια τέτοια αμνία στις εμπορικές συμφωνίες ε, της προνομιακής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, έχω μιλήσει με Αμερικανούς εκπροσώπους στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Νομίζω ότι και στην Ευρώπη υπάρχουν εκκρεμότητες. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε και εσείς κύριε Βότσον ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Point number eight. Περνάμε σημείο παριθμών 8. Η κυρία Βαϊντέρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή είναι ένα μέσο εξωτερικής πολιτικής που ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 για να δοθεί ε, βοήθεια σε τρίτες χώρες που έχουν ε, δυσκολίες προσωρινές όσον αφορά το ισοζυγείο πληρωμών. Βεβαίω αφορά χώρες οι οποίες ε, είναι ή θα μπορούσαν να είναι υποψήφιες, καθώς και κάποιες άλλες ε, της Κεντρικής Ασίας πλην του, της και του Τατζικιστάν. Συνολικά το ποσό που έχει δοθεί είναι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεις και δάνεια ή ε, ένας συνδυασμός και των δύο η βεβαίως γίνεται μετά από αποφάσεις κατά περίπτωση μια χρονοβόρα διαδικασία που έχει αντιμετωπίσει ε, πολλές επικρίσεις καθώς δεν είναι δυνατόν να δώσουμε τα λεφτά όταν χρειάζονται και είναι πιο επίγουσες οι ανάγκες μετά τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για μια πιο αποτελεσματική διαδικασία η Κομισιόν ε, προχώρησε σε κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές για την μακροοικονομική χρηματοδοτική σύνδρομη. Το έγγραφο είναι καλό, αλλά έχω καταθέσει κάποιε τροπολογίε. Θα προσπαθήσω να τι εξηγήσω σύντομα. Πρώτα απ' όλα, ο ορισμό τη ε, επιλέξιμη χώρα. Εγώ έχω αναφέρει χώρε υποψήφιε, ε, δυνητικά υποψήφιε και ε, χώρες της γειτονίας και έβγαλα τις ε, στρατηγικά σημαντικές χώρες, καθώς δεν είναι συγκεκριμένο και θα μπορούσε να καλύπτει οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Και έτσι θα μειώνονταν η διαθεσιμότητα της ε, συνδρομής ε, στις χώρες που προανέφερα, καθώς η χρηματοδότηση είναι πλέον μικρότερη σε σχέση με άλλα μέσα χρηματοδότησης της Ένωσης. Μιλάμε για 0,7 δισεκατομμύρια για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013. Κατόπιν ε, η νομοθετική διαδικασία υποστήριξε την πρόταση της Κομισιόν να αντικατασταθεί το υφιστάμενο σύστημα με την επιτροπολογία ε, και άρα θα υποβάλλεται μια πρόταση της Κομισιόν σε μια Επιτροπή Εκπροσώπων των Κρατών Μελών για να υιοθετηθεί με ειδική πλειοψηφία ως ε, μια ε, εφαρμοστική διάταξη. Παρά το ότι έτσι αποκλείεται το Κοινοβούλιο, είναι ο μόνος τρόπος να γίνει το μέσο αυτό πιο αποτελεσματικό και να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων. Εάν εισφαλίσουμε πως θα υπάρχουν σαφή και ακριβή κριτήρια για κατανομή των κονδυλίων αυτών, θεωρώ πως δεν θα υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα. Επιπλέον, σημειώνοντας πως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται κάποια εξαίρεση, πρότεινα σε εξαιρετικέ και αιτιολογημένε περιπτώσεις μια τρίτη χώρα μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη για το μέσο αυτό, αλλά στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να το κρίνουμε κατά περίπτωση με πράξη κατεξιοδότηση, με την επίσημη τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ ή κατά αυτά στο νέο άρθρο 11α. Επιπλέον έχω καθορίσει τον ρόλο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης συγκεκριμένα μέσω διαβουλεύσεων και αποφάσεων, παραδείγματο χάρη για την αναστολή των κονδυλίων και τακτικών ε, επανεξετάσεων, όπου πρέπει να ενημερώνονται εξίσου Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Η πρόταση τη Κομισιόν δεν ε, έκανε αναφορά στην υπηρεσία εξωτερική δράση, παρά το ότι πρόκειται για ένα μέσο εξωτερική πολιτική και τα κριτήρια επιλεξιμότητα επίση καλύπτουν και σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, δημοκρατίας και τα λοιπά. Ως αποτέλεσμα ήταν κάπως μπερδεμένη η διαδικασία, ενώ τα ζητήματα επιλεξιμότητας αναφέρονταν σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Τα άρθρα περί εκταμίευσης δεν τα ανέφεραν αυτά τα κριτήρια. Τέλος, με την πρόταση της ε, Κομισιόν, οι αλλαγές αυτές στις γενικές διατάξεις για την ε, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ε, θα έλεγαν 31 ε, Δεκάτου του 2013. Αυτό δεν είναι λογικό γιατί πιθανότατα θα υιοθετηθούν μόλις στο δεύτερο εξάμεινο του έτους αυτού. Θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να εφαρμοστούν οι αλλαγές αυτές ε, του κανονισμού στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο με μια επανεξέταση της εφαρμογής τους που θα υποβάλει η Κομισιόν σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και θα συνοδεύεται, αν είναι απαραίτητο, από νομοθετικές προτάσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες έχετε το σχέδιο της γνωμοδότησης και βεβαίω πάντα είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Άννα um, I, um... Εγώ είμαι ευγνώμων στη συνάδελφο Βάιδαρα για την εργασία της και τις επεξηγήσεις που μας έδωσε. Πιστεύω ότι πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των μελών σε αυτόν τον κανονισμό, διότι θα ήθελα η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας να είναι πιο ουσιαστική, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με τεράστιες ε, επιπτώσεις. Λέει εδώ ότι το σύστημα που προτείνεται είναι οικονομικά, γεωγραφικά και οικονομικά κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να είμαστε νομίζω πιο συγκεκριμένοι. σε σχέση με τις αρχές που θα πρέπει να καθοδηγούν την Ένωση σε σχέση με την οικονομική βοήθεια προς κάποιους εταίρους. βασικές αρχές όπως το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση της ε, διαφθοράς, αλλά και απασχόληση και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή η αίσθηση του ότι ασχολούμαστε μόνο με εσωτερικά θέματα, αντιμετωπίζουμε την κρίση, δεν είναι η σωστή αυτή η αίσθηση που δίνεται, αλλά μπας περιπτώσει είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό το κείμενο, θα το ξανακοιτάξω και θα το συζητήσω και με την εισηγήτρια. Ελπίζω να τραβήξει την προσοχή όλων των συναδέλφων γιατί και στο θέμα των κατεξοδότηση πράξεων Νομίζω πως θα έχει νόημα να εξασφαλίσουμε την ταχεία φύση της διαδικασίας. Να... Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα συμμετέχει με κάποιο τρόπο και το Κοινοβούλιο. Βλέπω πως έχουμε κάποιες μέρες μέχρι τα τέλη Μαρτίου να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Είναι ένας τομέας όπου πιστεύω πως η Επιτροπή μας θα πρέπει πραγματικά να δουλέψει και όχι να ικανοποιείται με κάποιες ε, τεχνικές ε, προτάσεις. Είναι πολιτικό θέμα. Κύριος Μαυρονικόλας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι η αντιμετώπιση τέτοιων δημοσιονομικών καταστάσεων χρειάζεται ένα εργαλείο αντιμετώπισης των κρίσεων που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Γι' αυτόν τον λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι πιο διαφανής και ειδικά σε νομικά ζητήματα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων να αποφεύγει χρονοβόρες διαδικασίες και καθυστερήσεις. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την αποδέχτρια χώρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του κανονισμού η σοσιαλιστική ομάδα, όπως ανάφερε και προηγούμενα η Άννα Γκόμες, τάσσεται υπέρ της οικονομικής βοήθειας τρίτων χωρών που δεν είναι απαραίτητα είτε υποψήφιες είτε ενδυνάμει υποψήφιες χώρες ή χώρες καλυπτώμενοι από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Το συγκεκριμένο εργαλείο χρηματοδοτικής συνδρομής χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται καμία χώρα ε, που βρίσκεται σε έκτακτη κρίση και χρειάζεται χρηματοδοτική συνδρομή για να αντεπεξέλθει. Επιπρόσθετα, η Σοσιαλιστική Ομάδα πιστεύει ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά και με αποτελεσματικό τρόπο στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην εφαρμογή τους όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης στην εκάστοτε χώρα θα αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ της αποδέχτριας χώρας, της Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση ανταπόκριση και αντίδραση από πλευράς της Ένωσης. Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει και έλεγχος για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Βαϊντέρε για την γνωμοδότησή της και συμμερίζομαι πολλά σημεία. Είμαι ο εισηγητής της ΣΥΝΤΑ για το θέμα αυτό και η έκθεσή μου ε, είναι παρεμφερής. Θα ήθελα και εγώ να εξασφαλίσω ότι η χρηματοδοτική συνδρομή ευθυγραμμίζεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας και εξασφαλίζει συνοχή των, των, της συνδρομής με την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να δίνεται χρηματοδοτική συνδρομή χωρίς να υλοποιούνται και να συντρέχουν τα κριτήρια των δημοκρατικών αρχών. Όπως και η κυρία Βαϊντέρε, και εγώ έχω επιμείνει στον ισχυρό ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης γιατί για το, την εξακρίβωση της επιλεξιμότητας κάθε χώρας ε, με βάση την σωστή εφαρμογή των δημοκρατικών μηχανισμών στη χώρα αυτή καθώς και στην ε, διαμόρφωση κάποιων μέτρων πολιτικής στα πλαίσια του Μνημονίου Συνανόησης. Είναι σημαντικό η ΕΕ να διαδραματίζει αυτό το ρόλο και συμφωνώ με τις τροπολογίες της κυρίας Βαϊντέρα. Σε ό,τι φορά την κάλυψη αναχώρα, η κυρία Βαϊντέρα πρότεινε κατά εξουσιοδότηση πράξης για την τρίτη κατηγορία των χωρών, που δεν είναι ούτε υποψήφιες ούτε χώρες της πολιτικής γειτονίας, αλλά από πολιτική, οικονομική και γεωγραφική άποψη βρίσκονται πλησίων της Ένωσης. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι δημοκρατίες Κεντρικής Ασίας συμπεριλαμβάνονται και Στη δική μου έκθεση εγώ προτείνω απλώς να προσθέσουμε τις ε, δημοκρατίες αυτές στη τρίτη κατηγορία των χωρών. Επίσης ε, θα πρέπει να προασπίσουμε και τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εξουσίες του. Οι περιπτωσιολογικές αποφάσεις, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνονται με εφαρμοστικές ε, πράξεις προκειμένου να επιταχυνθεί η χρονοβόρα διαδικασία λήψη αποφάσεων. Δεν συμφωνώ με την πρόταση αυτή γιατί ισχύει συναπόφαση για όλες τις ε, ε, προτάσεις μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Ε, γι' αυτό προτείνω κατεξουδότηση πράξης για κάθε περίπτωση χωριστά, με βάση τις νέες αρμοδιότητες που μας αναθέτει η συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι θα μπορέσουμε να ασκήσουμε αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και να γίνει το, το εργαλείο αυτό πιο αποτελεσματικό όπως επιθυμούν και οι ενδιαφερόμενοι. Αυτά και ευχαριστώ την κυρία Βαϊντέρη για την ανεκτήμητη της συνδρομή. Ευχαριστούμε, αγαπητέ συνάδελφε. Τώρα, οι τροπολογίες θα καταδοθούν μέχρι τις 29 Μαρτίου. 24 ε, Απριλίου ψηφοφορία στην Επιτροπή. Ε, έχουμε καθυστερήσει. 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα πολύτιμα σχόλιά σας. Ε, ήταν ανάλογα με αυτά τα οποία θα πρότεινα για να επιταχυνθεί η διαδικασία, να γίνει αποτελεσματική και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε το εάν το Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει το ρόλο του σε κάθε περίπτωση ή μπορεί να τεθούν κάποια κριτήρια που ανέφερε η κυρία Γκόμες. για να γίνει πιο αποτελεσματική διαδικασία βασιζόμενη στην Κομισιόν. Συμφωνώ πλήρω και το είπα και στην αρχή πω η υπηρεσία εξωτερική δράση πρέπει να παίξει ένα ρόλο, γιατί πρόκειται για ε, μια υπηρεσία που είναι πολύ ενήμερη για το τι γίνεται στις χώρες και ε, πρέπει να ενημερωνόμαστε και εμείς ως Επιτροπή ταυτόχρονα. Θα ήθελα να τονίσω πως ε, πρόκειται για ένα μικρό μέσο σε σχέση με άλλα και στόχο έχει να δει τις ανισορροπίες στα ισοζυγεία πληρωμών. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ για τα πολύτιμα σχόλιά σας και θα αρχίσω βεβαίως να εξετάζω τις ε, τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Εδώ και πέντε λεπτά περιμένει ο Υπουργός Εξωτερικών της Σομαλίας έξω από την πόρτα. Από την άλλη μεριά έχουμε βεβαίως ε, Έχετε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά και μόνο, κυρία Μακουβέη, γιατί βεβαίω χρόνο χρόνος δεν επαρκεί. Διαβάσατε φαντάζομαι την έκθεση αυτή για την Επιτροπή τη κοινοβουλευτική συνεργασία του Στις 16 Μαρτίου, πριν από λίγε μέρες μόλις, η Μολδαβική Βουλή εξέλεξε τελικά τον πρόεδρο και έτσι ξεπεράστηκε το σταγματικό αδιέξοδο. Ε, ο εκλεγμένος πρόεδρος είναι, ήταν προεδικαστή για πολλά χρόνια και ήταν και πρόεδρος ε, του Δικαστικού Συμβουλίου της Μολδαβίας. Κατάφεραν να, ε, να αποσπάσουν και τρεις ψήφους από τους κομμουνιστές και έτσι οι κομμουνιστές, τρεις κομμουνιστές συμφώνησαν με τους σοσιαλιστές ε, και ψήφισαν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωσής. Για την υπερδυνιστερία, πρόσφατες εξελίξεις. Από πέρυσι το Δεκέμβριο Έχουμε νέο πρόεδρο, δεν είναι ο κύριος Μπίγκροφ πια, και στο Βίλνιους έγινε ο πρώτος επίσημος γύρος στο διαπραγματεύσεως 5 συν και γίνονται πολλές επίσημες διαβουλεύσεις τις τελευταίες μέρες μεταξύ του Φιλάτ και του Προέδρου της Υπερδυστερίας. Υπάρχουν αναφορές για αυθαίρετες απαγωγές, κρατήσεις και φυλακίσεις από τις αρχές της υπερβριστερίας επίσης. Ευχαριστώ. Η εκλογή του νέου Προέδρου είναι πολύ χαρμό συνείδηση. Ελπίζω η κατάσταση να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό, η αμαλότητα Ευχαριστώ και θα προσκαλέσουμε τώρα τον Υπουργό Εξωτερικών της Σομαλίας. Ευχαριστώ. Kolleginnen und Kollegen, ich darf in unserer Mitte den Außenminister. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω τον Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνού Συνεργασία της Μαλιλάντ, η οποία συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταπολέμηση της πειρατείας και οπωσδήποτε μας απασχόλησε αυτό χτες και θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα για την κατάσταση στη Σομαλία συνολικά και στην ε, δική σας χώρα καθώς και το τι φαντάζεστε για περισσότερη σταθερότητα στην ε, περιοχή και την καταπολέμηση της φυρετίας Έχουμε και μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι λοιπόν για το ότι καταφέρατε να έρθετε εδώ πέρα γιατί ήσασταν και στη διάσκεψη του Λονδίνου για το μέλλον της ε, Σομαλίας. Φαντάζομαι πως είστε εξοικειωμένος με τον Πενελούξ. Γενικά είχατε ζήσει 12 χρόνια στην Ολλανδία και μετά 11 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κάνατε διδακτορικό στις ε, πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιχαμ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθατε εδώ πέρα και σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ε, για την Σομαλιλάνδη. Η χώρα μου έχει παλαιούς δεσμούς με την Ευρώπη και καλωσορίζουμε τις ε, σχέσεις αυτές και το ότι βεβαίως έχουμε ε, σχέση με πολλά κράτη-μέλη. Τα υφιστάμενα σύνορά μας είναι αποτέλεσμα της απεικιοκρατίας και του 19ου αιώνα. Μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία περάσαμε ε, στην Βρετανική Αυτοκρατορία και ενωθήκαμε θελοντικά με τη Σομαλία το 1960 και είχαμε κάποια ελευθερία. Η Ένωση βεβαίως δεν μας ωφέλησε ούτε μας ούτε τη Σομαλία και είχαμε μια ανεπιτυχή ε, συνεργασία. Τελευταίως είχαμε πολέμους ε, και αποδεκατίστηκε έτσι η πρωτεύουσά μας, ε, η Χαργέισα οι ηγέτες, μου, οι λοιπόν της ε, χώρας μου και της Σομαλίας συναντήθηκαν το 1991 και ανακήρυξαν ξανά την ανεξαρτησία μας και έκτοτε λειτουργούμε ως ανεξάρτητη χώρα αλλά αναμένουμε ακόμα ε, την διεθνή πολιτική αναγνώριση. Οι δύο δεκαετίες που ακολούθησαν από το 1991 μέχρι σήμερα ε, οδήγησαν σε δημοκρατική και ειρηνική Σομαλιλάνδη μέσω μιας δύσκολης διαδικασίας συμφιλίωσης σε τοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα κατέρευσε η κυβέρνηση στη Σομαλία και είχαμε τα προβλήματα που γνωρίζετε στο κέρας της Αφρικής. Τρομοκρατία, πειρατεία και πείνα. Οι προσπάθειε τη διεθνού κοινότητα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά δεν ήταν επιτυχημένε παρά τις ε, θυσίες που είχαν κάνει τα στρατεύματα της Αφρικανικής Ένωσης και τους πόρους που αφιέρωσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Στη Σομαλιλάνδη εμείς ε, ασχοληθήκαμε με την οικοδόμηση του δικού μας κράτους ε, με το να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας, χερσαία και θαλάσσια, να μην αφήσουμε τους πειρατέ να δράσουν από το εδαφός μας, να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και να έχουμε εσωτερικές δομές και να επιτρέψουμε στα 3,5 εκατομμύρια πολίτε μας να ζουν ειρηνικά και με ευημερία. Είμαστε υπερήφανοι για το ότι η Σομαλιλάδη λειτουργεί δημοκρατικά. Είχαμε πολλές διεθνές, ε, ε, πολλού διεθνείς παρατηρητές στις εκλογέ μας ε, και στις εκλογέ του 2010 που κατέληξαν σε ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας από το κόμμα που έχασε σε αυτό το οποίο νίκησε. Πρόσφατα λοιπόν άρχισαν ξανά επαφές με την διεθνή κοινότητα για να παίξουμε έναν ε, ρόλο στις ε, προκλήσεις που υπάρχουν στη γειτονική μας Σομαλία. Το προηγούμενο μήνα στην διάσκεψη του Λονδίνου, ο πρόεδρος τη χώρα μας και εγώ ως ε, υπουργό Εξωτερικών για πρώτη φορά παρευρεθήκαμε σε μια διάσκεψη για τη Σομαλία. Και νομίζω πως ε, αυτό ήταν ένα σημαντικό ορόσημο στην ε, διπλωματία μας. Ήμασταν ισότιμο μέρος της ε, διάσκεψης ε, και ο πρόεδρος ε, απίφθινε μια ομιλία προς το συνέδριο. Θεωρούμε ο πρόεδρος μας ο Αχμέντ Σιλάνιο. Θεωρούμε λοιπόν πως η λεγόμενη εδαφική ενότητα την οποία ζητάει η Σομαλία θέτει σε κίνδυνο την σταθερότητα την οποία έχουμε επιτύχει και αγνοείται έτσι η πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί επί τόπου καθώς είναι πολύ αποκεντρωμένη η πολιτική ε, σκηνή της, ε, των δύο χωρών. Και άρα θεωρούμε πως η ειρήνη και η σταθερότητα στο κέρας Αφρικής μπορεί να βαστεί κυρίως στην επιτυχία της ε, Σομαλιλάνδης. Αποτελούμε ένα σημαντικό παράδειγμα ειρήνης και δημοκρατική οικοδόμησης μιας χώρας από κάτω προς τα πάνω, βασιζόμενοι σε δοκιμασμένες μεθόδους στη χώρα μας για να μην υπάρχουν διαμάχες μεταξύ διαφόρων ε, φίλων. Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας, αυτή ακριβώς είναι η διαδικασία που έλαβε η χώρα στη Σομαλιλάνδη. Θεωρούμε πως μια παρόμοια προσέγγιση χρειάζεται και στη Σομαλία και προσφερθήκαμε να δώσουμε την εμπειρία μας του, στους αδελφούς μας στην Σομαλία και η Ευρώπη έχει τέτοια εμπειρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μια ένωση κρατών, αλλά και μια ένωση λαών. Δεν χρειάζεται να τονίσω στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών και την ε, δημιουργία κοινότητας από κάτω προς τα πάνω και το πόσο ε, θεμελιώδης είναι για ένα δημοκρατικό σύστημα παραδόσεις ε, σχεδόν καταστράφηκαν στη Σομαλία όσο μας ε, κυβερνούσε από το Μογκαντήσου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε σχεδόν το μισό κόστος των εκλογών μας του 2010 και έδωσε επίσης και οικονομική και τεχνική στήριξη ε, στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα της χώρας. Είναι η άποψη της κυβέρνησής μου και του λαού μας πως ο Μαριλάνδη θα ήταν σε ακόμη καλύτερη θέση να συνεισφέρει ε, σε μια ελεύθερη και σταθερή Σομαλία εάν ε, αναγνωριζόταν η χώρα μας ε, διεθνώς. Με μια τέτοια διεθνή αναγνώριση η Σομαλιλάνδη θα είχε πρόσβαση στις αγορές, στο διεθνές εμπόριο, στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα όργανα του. Οι περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις θα μας έδινε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε και σε διεθνείς οργανισμούς. Το ανακοινοθέν της διάσκεψης του Λονδίνου τον προηγούμενο μήνα αναγνώρισε και αναφέρω εδώ πέρα την ανάγκη να στηρίξουμε οποιοδήποτε διάλογο μεταξύ Σομαλάνδης και μεταβατικής κυβέρνησης του Μογκαντήσου για να ξεκαθαρίσουν τις μελλοντικέ τους σχέσεις. Αυτή η σαφής δήλωση ενισχύει την θέση μας για δύο χωριστές ε, οντότητες οι οποίες θα ξεκινήσουν έναν διάλογο ως ίσες για να δούμε τις μελλοντικέ μας σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στην αποδοχή του ότι η εθελοντική ένωση του 1960 μεταξύ Σομαλίας και Σομαλιλάνδης έχει αποτύχει και πως το μέλλον και η σταθερότητα και η ανάπτυξη των δύο χωρών μας εξυπηρετείται καλύτερα με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Σομαλιλάνδης. Έτσι θα μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη πολιτική ε, σταθερότητα την οποία χρειάζεται. Είμαστε σε επαφή με την διεθνή κοινότητα για την καταπολέμηση της πειρατείας ε, και της ε, τρομοκρατίας. Έχουμε ηγετικό ρόλο. Έχουμε περάσει ένα νόμο κατά της πειρατείας που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην περιοχή μας και επίσης άλλη σχετική νομοθεσία, ενδείξεις ε, που δείχνουν πως χώρα μας είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα, ειδικά με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταπολέμηση της πειρατεία και έχουμε θετικό ιστορικό και θα μπορέσω ίσως να επεκταθώ στην, ε, στη δευτερολογία μου. να ε, εκφράσω και πάλι την ευγνωμοσύνη μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για την συνεχιζόμενη στήριξη της ε, Σομαλιλάνδης. Ε, συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της είναι ο μεγαλύτερος δωρητής προς την χώρα μας, κάτι το οποίο εκτιμούμε πάρα πολύ και θα έλεγα πως η κοινωνία μας δεν θα μπορούσε να έχει επιζήσει χωρίς την στήριξη που της ΕΡΟΣΗ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα την ευχαρίστηση να συναντηθώ με τον Επίτροπο τον κύριο Πίμπαλξ, τον Επίτροπο Διεθνούς Ανάπτυξης, τον Ιούλιο του 2011. και ευκαιρία να συναντηθώ με υπουργού ανάπτυξης πολλών ευρωπαϊκών χωρών, Ολλανδίας, Βρετανίας, ε, Δανίας, που επισκέφθηκαν τη χώρα μας το τελευταίο 1,5 έτος. Ο πρόεδρος μας, ο Αχμέτ Σιλάνη, συνάντησε αρκετούς υπουργούς εξωτερικών της Ένωσης στο περιθώριο της διάσκεψης του Λονδίνου και αναμένουμε την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών μας με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Θα ήθελα λοιπόν να προσκαλέσω τους Ευρωπαίους Υπουργούς και Ευρωβουλευτές να επισκεφτούν τη Σομαλιλάνδη τους επόμενους μήνες για να μπορέσετε να δείτε από μόνοι σας ε, τα αποτελέσματα της γενεοδορίας της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, στις προσπάθειές μας να επιτύχουμε τους ε, στόχους ανάπτυξης χιλιετίας. Είτε στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης είτε της διοίκησης, η στήριξή σας παίζει ένα θετικό ρόλο στην ειρήνη και σταθερότητα και φόρα ανάπτυξη στη χώρα μου. Παραδείγματο χάρη, 19 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για να ανακατασκευαστεί η υποδομή ίδρευσης ε, στη χώρα μου. Επίσης ε, ε, προγράμματα εκπαίδευσης οδήγησαν στον ρυθμό παρακολούθησης του σχολείου να ανέβει από το 16% σε πάνω από 60% και καταφέραμε έτσι να γίνει δωρεάν η υποχρεωτική εκπαίδευση στην χώρα μου και να αυξηθεί η πρόσβαση ειδικά των κοριτσιών. Τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης βοήθησαν την ε, βελτίωση της αστυνομίας, των δικαστηρίων, ε, της κοινωνίας των πολιτών, της εκλογικής διαδικασίας και των συστημάτων οικονομικής διαχείρισης. Επίσης, ε, σημειώνω με ευχαρίστηση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα έχει αφιερώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για μια μελέτη σκοπιμότητας για τον διάδοχο Ντέρμπρα, από το λιμάνι δηλαδή Ντέρμπρα στην ενδοχώρα για να αυξηθεί η δυναμικότητα του λιμανιού αυτού και οι προοπτικές της χώρας μας. Το έργο αυτό βεβαίως έχει καθυστερήσει λίγο και χαρήκαμε ιδιαίτερα για το ότι τώρα προχωράμε στο... στην πάρα πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, η Σομαλιλάνδη θέλει να παίξει τον ρόλο τη στο να βρεθούν λύσει στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εκτιμούμε τι προσπάθειέ σα και μπορεί να γίνουν ακόμη περισσότερα πράγματα. Συγκεκριμένα, πολιτική αναγνώριση της Σομαλιλάνδης ε, ε, εντό των συνόρων που ορίστηκαν από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις τον 19ο αιώνα θα ενίσχυαν το ρόλο της ε, χώρας μας και έτσι θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικό εταίρο για την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα. Αντιλαμβάνομαι πως ο πρόεδρος του Νοτίου Σουδάν θα μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Θέλω να τονίσω πως έχουμε καλές σχέσεις με την κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν. Μάλιστα και ο πρόεδρός μας και εγώ ήμασταν επίσημοι προσκεκλημένοι του πρόεδρου Φαχίρε στην ορκομοσία του. Και έχουμε εμπορικές ε, σχέσεις και συνεργασία ασφαλείας με τον Νότιο Σουδάν. Ένα τελευταίο θέμα για την Αλσαμπάπ. Αντιλαμβάνομαι και είμαι σίγουρος πως ξέρετε πως ε, η Αλσαμπάπ ε, έχει σχεδόν ιτηθεί γύρω από το Μογκαντήσου με τη σχέση με την στήριξη των στρατευμάτων της Αφρικανικής Ένωσης. Αλλά το θέμα είναι πού θα πάνε αυτοί. Πού θα πάει η Al-Shabaab. Δεν νομίζω πως έχουν εξοντωθεί όλοι. Μόλις φύγουν από το Μογκαντήσου μπορεί να κατευθυνθούν προς Βοράν και αν πάνε στο ανατολικό κομμάτι της χώρας μας όπου υπάρχουν βουνά δύσκολα θα τους αντιμετωπίσουμε. Θέλω απλά να το τονίσω αυτό πως ο Μαλιλάνδη ε, πρέπει να στηριχθεί σε ζητήματα ασφαλείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας ε, σε έργα ανάπτυξη, σε εκπαίδευση υγεία, αλλά θα θέλαμε να έχουμε και συνεργασία για ζητήματα ασφαλείας. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τέτοια συνεργασία και θεωρώ πως ε, θα θέλαμε το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, οφθήσει και την Αφρικανική Ένωση να μας βοηθήσει. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση, υποδομές ε, στις δυνάμεις ασφαλείας. Μπορέσαμε να υπερασπιστούμε την δημοκρατία μας και την ασφαλεία μας εδώ και 20 χρόνια κατά των ακραίων και τζιχαντιστών ντόπιων και διεθνών. Αλλά δεν μπορούμε να πολεμήσουμε την al και την Al-Qaeda και τέτοιες ομάδες εάν ε, ανέβουν προς ε, Σομαλιλάνδη. Είμαστε ειδικά ευάλωτοι γιατί είμαστε δημοκρατική χώρα και οι αξίες που έχουμε δεν ε, είναι ιδιαίτερα αγαπητές τους ακραίους. Δεν θεωρούν πως η δημοκρατία, η ισότητα των φύλων, η ελευθερία έκφρασης είναι κάτι το θετικό. Γι' αυτό κινδυνεύουμε ιδιαίτερα λόγω των αξιών αυτών που εκπροσωπούμε και θα θέλαμε πολύ στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να σας πω πως, μια που αναφέρατε πως ε, ε, θα μιλήσει εδώ πέρα ο πρόεδρος του Νοτιού Σουδάν, αρρώστησε και τελικά δεν θα μπορέσει να, να παρευρεθεί. Τον λόγο έχει ο κύριος Γκάλερ. Να ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Στην Επιτροπή μας σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας είπατε. Θεωρώ πως είναι θετικό αυτό το οποίο μας λέτε πως η Σομαλιλάνδη υπάρχει και λειτουργεί ουσιαστικά ως κράτος εδώ και πολλά χρόνια και πως έχετε οργανωθεί με τρόπο δημοκρατικό και πως έχετε αναλάβει και αγώνα κατά της πειρατείας. Όταν λέω στο κομμάτι αυτό της Σομαλίας, ε, δεν εννοώ πως ε, ε, είμαι υπέρ του status quo φανατικά. Ούτως ή άλλως στην Ευρώπη τα τελευταία 22 χρόνια είδαμε πολλές αλλαγές των συνόρων η αρχή δηλαδή πως μπορούν να αλλάξουν τα σύνορα και να δημιουργηθούν νέα κράτη είναι κάτι το γνωστό στην Ευρώπη. Ως πρόεδρος ε, αντιπροσωπείας ε, για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο γνωρίζω πως παραδοσιακά μέχρι τώρα στην Αφρική η, η τάση αλλαγής των συνόρων ήταν περιορισμένη, αλλά ειδικά στην περιοχή σας, ειδικά με τον Νότιο Σουδάν, ε, υπάρχει ένα προηγούμενο ε, που ε, γίναν αποδεκτές οι πραγματικότητες. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω είναι πρώτον να συνεχιστεί η ρεαλιστική πολιτική, δηλαδή εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση de facto να συνεργαζόμαστε στον αναπτυξιακό τομέα να γίνονται έργα σε εσάς. χωρίς να ασχοληθούμε με το ζήτημα του στάτους του καθεστώτος. Αλλά η δεύτερη παράκληση είναι εσείς με τις δυνατότητές σας να συνεισφέρετε ε, έτσι ώστε στον νότο της χώρας να υπάρξει σταθερότητα Ακούσαμε χτες στην Υποεπιτροπή Ασφάλειας πως ε, υπάρχουν πολλά θετικά πράγματα στο Μογκαντήσου και Πέριξ, πως έχει νικηθεί ε, στην περιοχή του Μογκαντήσου η Σαμπάμπ και αποσύρεται. Η παράκλησή μου λοιπόν είναι να στηρίξετε αυτή την ε, διαδικασία και να μην ε, σκεφτείτε τακτικά και να συνάψετε έτσι συμμαχίες με ομάδες που ε, είναι αντίπαλοι αυτών ε, που δρώνουν στο Μογκαντήσου. Θα πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα μια σταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή του Μογκαντήσου και μετά το ζήτημα του καθεστώτος να ρυθμιστεί αργότερα και επισήμως. Όπως είπα, εγώ δεν θέλω να διατηρηθεί ένα τεχνητό status quo αιώνιος, όπως το χαρακτηρίσετε κι εσείς, αλλά δεν θέλω οι στόχοι που έχετε να πλήξουν άλλες θετικές εξελίξεις ε, στην ε, Σομαλία με ε, στόχο το καθεστώς το δικό σας. Αυτό είναι, αυτή είναι η παρακλησή μου και θα ήθελα να μάθω την άποψή σας. Καλώς ορίσατε, Υπουργέ. Και καλώς ορίζω τα όσα είπατε, γιατί έχουν νόημα, βγάζουν ένα νόημα. Και κυρίως γιατί όσο περισσότερο προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει στην Σομαλία, τόσο περισσότερο θυμώνω με τη συνανεπάρκεια των πολιτικών μας. Και δεν εννοώ μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τη διεθνή κοινότητα ως σύνολο. Πράγμα που έχει τεράστιες επιπτώσεις όσον αφορά το πόσο υποφέρει ο κόσμος, ο λαός της Σομαλίας, που είναι η προτεραιότητά μου. Τα όσα είπατε λοιπόν έχουν νόημα και εγώ ανέκαθεν ζητούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί μαζί σας και να μην βασίζεται μόνο σε αυτή τη DFG που είναι τελείως τεχνητή, τη μεταβατική κυβέρνηση που είναι τελείως τεχνητή. Και θα ήθελα Καταλαβαίνω βέβαια το αίτημα της ε, ανεξαρτησίας της Σομαλιλάνδης, αλλά βλέπετε ότι αυτή η μεταβατική κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι ένα συνομιλητής για το υπόλοιπο, αυτό που λέγεται Σομαλία, όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση της. Εγώ είμαι ευτυχής γιατί ως αποτέλεσμα της δέσκεψης του Λονδίνου υπάρχει αυτή η δέσμευση και η ε, επαφή με τη Σομαλιλάνδη την οποία περιγράψατε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για την Αφρικανική Ένωση που έχει έδρα στην διπλανή σας χώρα, την Αιθιόπια. Εσείς συνεργάζεστε με την ε, Αιθιοπία στο πλαίσιο της ε, ΑΓΙΑΝΤ. Αυτά είναι μηνύματα λοιπόν τα οποία μπορούν να περάσουν από τα κράτη της Αφρικανική Ένωση. Και ως προς αυτό κατανοούμε βεβαίως την απροθυμία η, ε, αποσύνθεση των υφιστάμενων συνόρων και κρατών, αλλά είδαμε επίσης τις εξελίξεις για τον Νότιο Σουδάν. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρξει κάποιο είδους κυβέρνηση σε αυτή την ε, χώρα, τη Σομαλία. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας ενημερώσετε για το, την Αφρικανική Ένωση και και για την Αιθιοπία. Ορισμένοι πιστεύουν πως οι Αμερικανοί πιέζουν την, πίεσαν την Αιθιοπία να εισβάλλει στην Σομαλία το 2006 και ήταν χειρότερη αυτή η συνταγή λόγω των όσων προκάλεσε και ποιος είναι ο ρόλος που παίζει τώρα η Αιθιοπία στο κέρας της Αφρικής. Και έπειτα, για το νόμο για, κατά της πειρατείας, έχω την εντύπωση πως ασχολούμεθα με την πειρατεία από την άποψη ορισμένων ε, ομάδων συμφερόντων εδώ, στην δική μας πλευρά του κόσμου, που δεν αντιπροσωπεύουν όμως και τα συμφέροντα των λαών της περιοχής σας. Νομίζετε πως αυτό, αυτή η εντολή κατά της πειρατείας ε, θα αποφύγει και τα εγκλήματα κατά του λαού σας ε, όσον αφορά τα ύδατα, τους πόρους, τους αλληλευτικούς, το περιβάλλον. Πράγματα που βρίσκονται σε αυτό, στη βάση αυτής της τόσο επικερδούς υπόθεσης της πειρατείας. Και επίσης, αν θα μπορούσατε να μας πείτε Ποια κατά τη γνώμη σας είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για να ιτηθεί ε, η Al-Shabaab σε ολόκληρη την περιοχή. Τάνοκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, εδώ βρίσκομαι. Σας καλωσορίζω και τον Μοχάμεντα, Αλ, ε, τον εκπρόσωπό σας που κάνει εξαίρετη δουλειά. Δεν χρειάζεται καμία εισαγωγή στην κυβέρνηση της Ομαλιλάνδης γνωρίζετε ότι είμαι υπέρ της επαναναγνώρισης της ανεξαρτησίας σας αναγνωρίστηκε το κράτος σας για μια εβδομάδα πριν μπείτε σε αυτή την ατυχή γάμο με την πρώην Ιταλική Σομαλία ε, ανάμεσα στο 60 και το 61. Πολλά παραδείγματα υπήρξαν ε, στην Αφρική και στην Μέση Ανατολή για γάμους που οδήγησαν σε διαζύγια και νομίζω πως το καθεστώς σας στο πλαίσιο διεθνούς, ε, διεθνής νομοθεσίας είναι πολύ ισχυρότερη η δική σας υπόθεση από ό,τι το κοσυφοπαίδιο για ανεξαρτησία. Εγώ ανέκαθεν θεωρούσα πως η αυτοδιάθεση είναι πολύ σημαντική και η εδαφική ακεραιότητα, αλλά όχι απόλυτες αρχές όσον αφορά τη δημιουργία ενός κράτους. Ωστόσο πιστεύω πως εσείς πληρείτε όλα, αν, τα περισσότερα αν όχι όλα, ε, τα κριτήρια, τα παραδοσιακά, ε, για να φτιάξετε το δικό σας κράτος και γιατί έχετε καταπολεμήσει και την τρομοκρατία με τη μορφή της Αλσαμπά και θα πρέπει φυσικά να σας βοηθήσουμε να καταπολεμήσετε την τρομοκρατία στη χώρα σας και στην Πούντλαντ και θα πρέπει να βρούμε και τα κονδύλια για να βοηθήσουμε να φτιάξετε νέες εγκαταστάσεις σοφρονιστικές για να φυλακίσετε τους πειρατές, γιατί δεν φτάνει μόνο να τους πιάσετε. Επίσης, εγώ ενθαρρύνθηκα πολύ από το τελευταίο ανακοινοθέν της διάσκεψης του Λονδίνου που αναφέρει τη Σομαλιλάνδη χωρίς να λέει λεπτομέρειες, αλλά δίνει ένα είδος πολιτικού όντως κάποιου είδους ε, υπάρχει μια καθυστερημένη αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα ότι η μεταβατική κυβέρνηση που φτάνει σε αυτή την, στο τέλος της άχρηστης ζωής της θα πρέπει να οδηγήσει στον προβληματισμό για το μέλλον της Ομαλιλάνδης και για το καθεστώς. Έχω Συμφωνώ με το αυτό που είπε ο κ. Γκάλλο, ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να εστιάσουμε στο καθεστώ, αλλά πάντω δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η κυβέρνηση, ο λαό σα, θέλετε βασικά αυτό που δόθηκε και στη Γαλλική Σομαλία, στο Τζιμπουτί, που θέλετε να γίνετε ανεξάρτητο κράτος, το Τζιμπουτί έγινε ανεξάρτητο, ε, είναι ευημερή, είναι ειρηνικό, έχει καλή συνεργασία. Αν ήσασταν ανεξάρτητο κράτος θα μπορούσατε να μπείτε σε ένα σωρό ρίς και περιφερειακές συνεργασίες με το Μογκαντήσου, με την Αιθιοπία, με οποιονδήποτε. Και θα πρέπει να πω ότι το έχω μελετήσει αυτό και για το θέμα της Αιθιοπίας. Νομίζω ότι η δράση της Αιθιοπίας στην περιορισμένη εισβολή στην Σομαλία βοήθησε γιατί εξ, ε, ε, εκρίζωσε την τρομοκρατία της Αλ Σαμπάμπα όπως και ε, στα νότια. Η Σομαλιλάνδη μόνη δεν μπορεί να τα καταφέρει και εγώ που είμαι εισηγητής για την έκθεση αυτού του κοινοβουλίου που θα εκπονηθεί στο μέλλον για το κέρας της Αφρικής θα εστιάσω σε όλα αυτά τα θέματα συμπεριλαμβανομένου του θέματος της Ομαλιλάνδης και του δικαιώματος για επανακαθορισμό όσον αφορά την δέσμευσή μας και την εντολή για τις διάφορες στρατιωτικές θαλάσσιες επιχειρήσεις που θα μπορούν να συνεχίζονται και στις ακτές της Σομαλίας ώστε να διώκουν τι εγκαταστάσεις των πειρατών. Ε, και μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση στη διάρκεια του μεσημεριανού γεύμα. Πάντως να είστε βέβαιοι ότι η ομάδα μου υποστηρίζει τη χώρα σας και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστήσουμε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην χώρα σας και ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζωτικά προγράμματα υποδομών που θα τα συζητήσουμε το μεσημέρι. Να μην μιλάτε για φαΐ... Γιατί εγώ δεν είμαι προσκεκλημένος. Ο κύριος ε, Κέλλαμ. Ευχαριστώ και σας ε, καλωσορίζω θερμά κύριε ε, Υπουργέ Εξωτερικών. Είμαι ε, από την Εσθονία. Νομίζω ότι η χώρα σας έχει πραγματοποιήσει πολύ εντυπωσιακή πρόοδο μετά την αναρχία και το διχασμό στην επικράτεια της γειτονικής σας χώρας. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι εσείς ήδη περάσατε το τεστ της ανεξαρτησίας, γιατί έχετε εξασφαλίσει κράτος δικαίου και σταθερότητα που είναι απαραίτητες αρχές. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Οι αιτίε της διαφοράς και του διαχωρισμού από τη γειτονική σας Σομαλία είναι εθνοτικές ή πολιτικές. Αναφερθήκατε στο διάλογο. Είπατε ότι είστε, πρόθυμος, είστε πρόθυμοι να έχετε διάλογο με τη Σομαλία. Ποια θα ήταν κατά τη γνώμη σας η ιδεώδης έκβαση ενός τέτοιου διαλόγου, μια στενότερη συνεργασία με τη χώρα αυτή. Και τέλος, για τα οικονομικά. Τι κλάδι της οικονομίας θα τραβήξουν το ενδιαφέρον σα σε τι θα επικεντρωθείτε τι γίνεται με την παιδεία στη χώρα σας. Μπορείτε να εξασφαλίσετε επαρκή ανώτερη παιδεία στους νέους ε, συμπατριώτες σας ή μήπως υπάρχει μια έξοδος, μια αποδημία των νερών. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την νεολαία του Ισομαλιλάνδης να παραμείνει και να σπουδάσει εκεί. Η κυρία Σβένσον, Ο κύριος Βένσον μάλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες που μας δώσατε κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι μας ενημερώσατε για την κατάσταση στη Σομαριλάνδη και θα ήθελα να εκφράσω τον αμέσω θαυμασμό μου για τη σταθεροποίηση που επιτύχατε, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις γειτονικές σας χώρες. Μας ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει κάτι που είπε και ο κύριος Κέλαμ ιδιαίτερος γίνεται στη σχέση σας με τις γειτονικές σας χώρες. Τι προπτικές ε, συνεργασίας και εξελίξεων υπάρχουν, γιατί η Σομαλιλάνδη εξαρτάται από τα αρδευτικά συστήματα, οπότε οι σχέσεις με, τη, με τους γείτονές σας ε, θα έχουν κεφαλαιώδη σημασία. Ποια είναι η γνώμη σας λοιπόν, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν οι σχέσεις σας με τις γειτονικές σας χώρες. Ο κύριος Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό μας για αυτά τα οποία έχετε επιτύχει στην πατρίδα σας τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκόμες, πως θα ήταν σημαντικό και για το μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί και να συνεργαστεί εντονότερα με περιφερειακούς παίκτες και να μην προσανατολιζόμαστε μόνο με τις αρχές του Μογκαντήσου. Παρ' όλα αυτά, τώρα έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ο κύριος Ρόντος, ο ειδικό απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήρθε εδώ πέρα χτες και μας είπε για το τι κάνει, για το ότι ο δικός χάρτης του Τζιμπουτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί ε, μέχρι τον Αύγουστο. Εμένα θα με ενδιέφερε να μάθω ποιο ρόλο βλέπετε εκεί πέρα για τη Σομαλιλάνδη. να σας πω πως ε, θεωρώ πως είναι στρατηγικό λάθος αντί να ε, λάβετε μέρος σε αυτή τη διαδικασία να θέσετε το ζήτημα της ανεξαρτησίας. Ανεξαρτησία υπάρχει σε πολλές μορφές. Στην πατρίδα μου παραδείγματο χάρη υπάρχει το ελεύθερο κράτος της Βαβαρίας όπως λέμε ή της Σαξονίας. Έχουν κρατική υπόσταση αλλά είναι μέλος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Αλλά αυτό είναι ζήτημα μακροπρόθεσμο. Τώρα όμως τίθεται το ζήτημα ε, το πώς θα ξεπεράσουμε την αστάθεια που υπάρχει και δεν μπορεί να είναι η ε, προοπτική να είναι η Σομαλιλάνδη ανεξάρτητη και να περικυκλώνεται από μια θάλασσα αστάθεια. Θα πρέπει λοιπόν να συνεισφέρεται νομίζω πρώτα απ' όλα στην επίτευξη της σταθερότητας. Εσείς ο ίδιος είπατε πως η Αλσαμπάμπ, ένας παράγοντας της αστάθειας, πιθανώς να προσπαθεί να επεκταθεί προς βορρά, προς Πούντλαντ ή και Σομαλιλάνδη. Είπατε πως θέλετε στήριξη. Νομίζω πως αυτό το ίδιο το οποίο ζητάτε ε, παραπέμπει στο τι πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε κάτι το ξεκάθαρο για τις προτεραιότητές σας. Κατόπιν μιλήσατε για αυξημένη στήριξη ασφαλείας. Τι συγκεκριμένα εννοείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. το κατά πόσο τώρα η μεταβατική κυβέρνηση είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής, κάτι που ρώτησε η κυρία Γκόμες. Η μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση συστήθηκε το 2004 στην Κένια και στόχο της είχε να διαχειριστεί και να υλοποιήσει κάποια μεταβατικά καθήκοντα, κυρίως τη διαδικασία επανασυμφιλίωσης επανασυμφιλίωση των πολιτικών φορέων σε ολόκληρη τη Σομαλία. Δεύτερο καθήκον, δεύτερη αποστολή της μεταβατικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης ήταν να τροποποιήσει το πολιτικό κατεστημένο, δηλαδή ε, να ε, ε σύνταγμα, να διοργανώσει εκλογές και να αναθέσει την εξουσία σε ένα εκλεγμένο σώμα. Επίσης, θέλει να εξασφαλίσει την ε, επαναφορά της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Σομαλία. Δυστυχώς απέτυχε στις αποστολές αυτές. Δεν κατάφερε να υλοποιήσει ούτε ένα από ε, τα καθήκοντα που είχε αναλάβει η μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Από το 2004 επαναλαμβάνω τότε που συστήθηκε. Έχουν περάσει 6-8 χρόνια. Ε, βέβαια κάθε φορά ζητούσαν παράταση της εντολής, με το που τελείωνε εντολή πήγαινα στο Τζιμπούτι την Καμπάλα ζητώντας παράταση της εντολής και του έργου. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι η μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι κατά ανάγκη ε, αξιόπιστος ε, συνομιλητής ή ικανή να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της περιοχής, γιατί τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Περαιτέρω ανάλυση είναι περιττή. Πάντως, η συμφωνία του Τζιμπουτή και η συμφωνία της Καμπάλα ουσιαστικά παρέτειναν την εντολή της μεταβατικής κυβέρνησης. Δεν προσδιορίσα διαφορετικό πλαίσιο για τη Σομαλία. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να παραταθεί περαιτέρω η εντολή της μεταβατικής κυβέρνησης. Συμφωνώ ε, ότι τον ε, Αύγουστο θα πρέπει να αποχωρήσει η μεταβατική κυβέρνηση και να δώσει τη θέση της, ε, να παραχωρήσει τη θέση σε μια νέα διοίκηση σε ό,τι αφορά την ε, σχέση Αφρικανικής Ένωσης και ε, σχέση μας με την Αιθιοπία. Συνεργαζόμαστε στενά με την Αιθιοπία, τον Τζιπουτή, την Κένια και θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας και στην Αφρικανική Ένωση. Αλλά δεν είμαστε επισήμως μέλος της Αφρικανικής Ένωσης. Ως εκ τούτου ε, επιδιώκουμε κάποιο ειδικό καθεστώς, έστω και παρατηρητή, ώστε να μπορέσουμε να εκφέρουμε τη γνώμη μας και σε διεθνή φόρα, όπως είναι αυτό της ε, Αφρικανικής Ένωσης ή της ε, ΑΙΚΑΤ, ούτε και εκεί είμαστε μέλος. Γι' αυτό ζητούμε από τα αφρικανικά κράτη να διευκολύνουν ε, την προσχώρησή μας σε τέτοια φόρα για να μπορέσουμε να εκφέρουμε εκεί τις απόψεις εμπειρίες και τις προσδοκίες μας. Η επέμβαση στη Σομαλία από γειτονικέ χώρες. Το 2006 έγινε μια επέμβαση στη Σομαλία μια εισβολή. Ε, νομίζω ότι το σομαλικό ζήτημα μόνο οι Σομαλοί είναι ικανοί να το επιλύσουν. Δεν θεωρούμε ότι ε, από όπου και προέρχονται οι επεμβάσεις εξωτερικές μπορούν να συμβάλλουν σταθερότητα. Βέβαια, η μεταβατική κυβέρνηση είναι εμφανώς αναποτελεσματική, ούτε καν το Μογκαντήσιο δεν μπορεί να εξασφαλίσει. Οπότε χρειάζεται μια διεθνή εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για παράδειγμα. Είναι καλή αυτή η πρόταση για παρουσία διεθνών δυνάμεων με διεθνή εντολή για να εξασφαλιστεί ένα είδος ασφάλειας εκεί. Αλλά για να διαιωνιστεί αυτή η ασφάλεια θα πρέπει να έχουμε ένα σομαλικό κράτος και να δοθεί ευκαιρία στους Σομαλούς να το διοικήσουν. Η δική μας ε, ασφάλεια και σταθερότητα απέρευσε από εμά του ίδιου, όχι από τι διεθνεί δυνάμει από εξωτερικέ ε, επεμβάσει. Και τώρα δρεύουμε του καρπού τη ειρήνη, τη σταθερότητα και τη ασφάλεια. Ε, βλέπουμε την οικονομική ανάπτυξη και βλέπει ο λαό μα, ο κόσμο μα, τα ωφέλη τη ε, ασφάλεια. Και φαντάζομαι ότι και στη Σομαλία δεν θα υπάρξει διαφορά. Σε ό,τι αφορά την πειρατεία, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε έναν νόμο κατά της πειρατείας αλλά το κατά πόσο οι διεθνείς ε, ε, επιχειρήσεις ήταν επιτυχείς. Νομίζω ότι αν ήταν επιτυχείς οι διεθνείς επιχειρήσεις θα είχε μειωθεί η πειρατεία, κάτι που δεν ισχύει ιδιαίτερος. Δεν ήταν τουλάχιστον τόσο επιτυχημένες όσο θα περιμέναμε αυτές οι διεθνείς επιχειρήσεις. Περιμένουμε μια πιο ολοκληρωμένη περιεκτική προσέγγιση για την καταπολέμηση της πειρατείας. Και το θέμα δεν είναι εδώ να έχουμε στρατεύματα ή ναυτικές δυνάμεις. Είναι να δώσουμε ευκαιρίες στους ε, νέους της Σομαλίας, ε, να ξαναφέρουμε τη σταθερότητα ε, στη Σομαλία, να αναλάβει μια κανονική κυβέρνηση, για να μπορέσει η Σομαλία μόνη της να προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα θα πρέπει η ίδια η Σομαλία να προσφέρει θέσει απασχόληση στους νέου στου πολίτε τη για να έχουν εναλλακτική λύση, να μην είναι υποχρεωμένοι να καταφεύγουν στην πειρατεία για να επιβιώσουν. Χρειαζόμαστε μια περιεκτική και ολιστική προσέγγιση, πέραν τη προσέγγιση με μοναδικό πρίσμα την ασφάλεια που υιοθέτησε η διεθνή κοινότητα για να καταπολεμήσει την πειρατεία. Διαχωρισμός, διαίρεση, διάλογος και ανάπτυξη της οικονομίας. Ο λαός της Ομαλιλάνδης ζήτησε να διατρανώσει ε, ε, την ε, ανεξαρτησία της. Εμείς δεν αποσχιστήκαμε. Διαλύθηκε μια ένωση. Επιβεβαιώσαμε την ανεξαρτησία μας. Ήμασταν και προηγουμένως ανεξάρτητο κράτος. Οικειοθελώς προσχωρήσαμε σε ένωση με τη Σομαλία και θελήσαμε να διαλύσουμε πια αυτή την ένωση. Το ίδιο συνέβη και με την Κάμπια. Κάποια στιγμή υπήρχε ένωση και κάποια στιγμή διάσπαση. Δεν ήταν απόσχηση ούτε αλλάζουμε τα σύνορα. Κανένα σύνορο δεν αλλάζουμε. Ήταν απικιακρατικά αυτά τα σύνορα. Εμείς δεν αλλάζουμε επιτόπου τα σύνορα. Επανερχόμαστε στα παλιά σύνορα, στα αρχικά σύνορα, όπως υπήρχαν και πριν την αύξηση των απικιακρατικών δυνάμεων και όπως διαμορφώθηκαν μετά. Δεν αλλάζουμε λοιπόν τα σύνορα, όπως κάνουν άλλες αποσχιστικές οντότητες ή χώρες. Οικονομική ανάπτυξη. Η αλληλεία είναι ένας κλάδος που μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε, γιατί έχουμε ε, υποεκμετάλλευση των χωρικών μας υδάτων. Δεν έχουμε καν την ικανότητα και την τεχνολογία για να αλλιεύσουμε στα υδατά μας, ούτε μπορούμε ούτε έχουμε τις εγκαταστάσεις ε, για μεταποίηση, κατάψυξη, προκειμένου να εξαγάγουμε τα αλληλευτικά μας προϊόντα, ούτε έχουμε εξαγωγικές ε, διεξόδους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διοχετεύσουμε τα αλληλευτικά μας προϊόντα. Επίσης έχουμε και ορυκτό πλούτο, έχουμε πετρέλαιο για παράδειγμα και εκεί θα θέλαμε να προσελκύσουμε ε, αλλοδαπές διεθνείς επενδύσεις. Και στο λιμάνι της Μπέρμπρα θα πρέπει να γίνει μια ανασυγκρότηση του λιμανιού γιατί νομίζω ότι θα εξυπηρετήσει το σύνολο του κέρατος της Αφρικής μια τέτοια αναβάθμιση του λιμανιού της Δέρμπρα. Ε, και χαίρομαι για το ενδιαφέρον που έδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, μελέτη, τη μελέτη που έγινε, η μελέτη της σκοπιμότητας και την ε, αναμόρφωση του λιμανιού της Δέρμπρα μας χαροποιεί ιδιαίτερος. Ο δικός χάρτης του Αυγούστου και το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Σομαλιλάνδη ως προς τη Σομαλία. Ο στόχος μας είναι σαφής, να γίνουμε κυρίαρχο ανεξάρτητο κράτος που θα αναγνωρίσει η διεθνή κοινότητα. Αυτό είναι ο στόχος μας. Βέβαια, μερικές φορές η υλοποίηση των στόχων χρειάζεται κάποιο χρόνο. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια, η ανάπτυξη, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ε, να παρέχουμε υπηρεσίες παιδεία υγεία στο λαό μα. Αυτό κάνουμε τα τελευταία 20 χρόνια και χάρη στου φίλου μα, όπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε, χάρη σε άλλε χώρε μπορούμε να προσφέρουμε αυτέ τις υπηρεσίε, Θέλουμε να τι αναβαθμίσουμε και να γίνουμε αξιόπιστοι, να δίνουμε την εντύπωση αξιόπιστη κυβέρνηση, όπω είπαν και οι ευρωβουλευτέ. Αυτή είναι η άμεση στόχη, οι άμεσε προτεραιότητές μα, Αλλά ο απότερο σκοπός μας είναι να γίνουμε κυρίαρχο ανεξάρτητο κράτος κυρίαρχο κράτος. Ο δικό χάρτη έχει αποτύχει. Δεν απέφερε καρπού. Φαίνεται ότι ε, το ανακοινωθέν τη διάσκεψη του Λονδίνου αντικατέστησε τον οδικό χάρτη που έδωσε ένα πλαίσιο για τη Σομαλία. Και η παράγραφος 6 του ανακοινωθέντος ε, λέει σαφώ ότι η Σομαλία και οι Σομαλιλάδοι μπορούν να τύχουν υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα αν συμφωνήσουν να καθίσουν σε μια τράπεζα των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν τις μελλοντικές σχέσεις. Εμείς πολύ ευχαρίστω να ε, συνομιλήσουμε με τη Σομαλία εφόσον αναλάβει μια αξιόπιστη κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να, να συνομιλούμε με μια ομάδα πολιτικών που έχουν ακόμη τρίμηνη θητεία. Εμείς ε, επιζητούμε την ε, διεθνή υποστήριξη και της Σομαλίας. Θέλουμε να συνεχίσετε να συνδράμετε τη Σομαλία. Θέλουμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες ε, και απόψεις με τη Σομαλία. Θέλουμε να διευκρινίσουμε τις σχέσεις μας. Θέλουμε να γίνουμε ανεξάρτητοι. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βοηθήσουμε τη Σομαλία και πιστεύω ότι με την ανεξαρτησία μας θα έχουμε μια πολύ καλύτερη ευκαιρία για να στηρίξουμε τη Σομαλία πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε γειτονική χώρα. Σας ευχαριστώ. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου. Herr Minister, herzlichen Dank für Ihre klaren Darlegungen. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για τις αφείς ε, δηλώσεις σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία για την σταθερότητα δηλαδή της χώρας σας, ε, την χρηστή διοίκηση και για να έχει η νεολαία της Ομαλιλάνδης προοπτικές όπως το περιγράψατε. Μου φαίνεται ότι είπατε τα σωστά και σημαντικότερα πράγματα και νομίζω πως θα έχετε και την υποστήριξη της Επιτροπής μας. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στο μόνο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, λέει τη